Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αφήσαμε το ακαδημαϊκό τέταρτο για λόγους ευγενίας, αλλά πρέπει να αρχίσουμε γιατί έχει έρθει υπουργό κ. Ζόλταν Μπάλοκ, Υπουργό Κοινωνική Ένταξη τη Ουγγρική Κυβέρνηση, για να μα παρουσιάσει τα συμπεράσματα τη Ουγγρική Προεδρία σχετικά με την κοινωνική ένταξη και ιδιαίτερο στην ένταξη των Ρωμά. Βεβαίω αποτελεί τιμή για μας η παρουσία του Υπουργού εδώ, καθώς εχθές ε, δεχτήκαμε τους Υπουργούς Αυρίσκη και τον Υπουργό Εστερικών, τον κύριο ε, Πίντερ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ, και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψαμε μου μητρική μου στα Ουγγρικά. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε, και κύριοι. Θα θυμάστε σίγουρα τον Ιανουάριο όταν είχα έρθει στην ακρόαση μου σας είπα στο τέλος της συνεδρίασης ότι θα έρθω να σας αναφέρω στο τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας για να σας πω πώς προχωρήσαμε στα σχέδιά μας και τι πετύχαμε. Αποτελεί λοιπόν ιδιαίτερη χαρά για μένα το γεγονός ότι πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει ως προς την ένταξη το Ρωμά. Έγιναν πολλές διαπραγματεύσεις, καθόλου εύκολες πρέπει να σας πω, το θέμα είναι πάρα πολύ ακαθόδες ευαίσθητο και λεπτό. Η ένταξη, το Ρωμά, ε, κοινωνική ένταξη δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση και τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 27 και χρειάστηκε να συνονοηθούν όλες οι χώρες. Πάντως η κατάσταση, ε, βέβαια πρέπει να σας πω, διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή και ε, σημεία θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς τη συνεργασία των οποίων δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις επιτυχίες. Επιτρέψτε μου να σας ε, μιλήσω για το εξάμεινο που μας πέρασε. Όπως σας ανέφερα ήδη τον Ιανουάριο, η κατάσταση των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας ανησυχεί. Η ομάδα αυτή του πληθυσμού ε, είναι ετερογενής. Συνολικά 8 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υφίστανται ε, διακρίσεις, υποφέρουν από ένδια και από ε, χωριστή αντιμετώπιση. Ασχολούνται κυβερνήσεις και, και μη κυβερνητικές οργανώσεις με το θέμα και τα προβλήματα των Ρωμά από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια δεν μπορεί κανείς να πει ότι γνωρίσαμε καμπή στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης στο Ρωμά. Η κοινωνική ένταξη στο Ρωμά στο Δινικές είναι κάτι το οποίο θεωρούμε αναπόφευκτο και πάρα πολύ σημαντικό και επιθυμητό. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη αλλά και πολλοί διεθνείς οργανισμοί τόνισαν την ανάγκη να ενταχθούν οι Ρωμά στις κοινωνίες μας. Και για την Ουγγαρία ήταν πολύ σημαντικό το θέμα και συνδεόταν και με κινδύνους. Για μας ε, λοιπόν αποτέλεσε στη στρατηγική μας ύψιστη προτεραιότητα. Στην Ουγγαρία η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι καθόλου ρόδινη. Στις 9 Μαρτίου εγκρίνεται ένα σχέδιο ψηφίσματος της κυρίας Λίβια Γιάροκα ε, με θέμα την ένταξη και την κοινωνική συμμετοχή των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Στη στρατηγική αυτή βλέπουμε σημαντικές προτάσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια στις 5 Απριλίου ενέκρινε μια ανακοίνωση για ένα σύστημα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 και σε, σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Τέσσερα είναι τα βασικά πεδία που έχουν εντοπιστεί εδώ. Παιδεία, στέγη, απασχόληση και υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε ε, τα κράτη-μέλη να ορίσουν και το οικονομικό πλαίσιο για να γίνουν πραγματικότητα αυτή η στόχη. 7 και 8 Απριλίου ακολούθησε στη Βουδαπέστη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής ε, Πλατφόρμας για τους Ρωμά. Η διοργάνωση ήταν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς το συνδέσαμε και με κοινωνικές εκδηλώσεις, με πολλούς καλλιτέχνες ε, Ρωμά, μουσικούς, ε, χορευτές, ε, τραγουδιστές. Και είχαν την ευκαιρία όλοι, όχι μόνο εκείνοι που συμμετείχαν στη διάσκεψη, να γνωρίσουν την κατάσταση, να γνωρίσουν και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δουν τις δράσεις της Προεδρίας. Επίσης, συστήσαμε εκεί και κάποιες θρησκευτικέ κοινότητες, εκτός από το πρόγραμμά μας. Ακολούθησαν και άλλες δράσεις, ε, το Συμβούλιο επιλήφθηκε του θέματος ε, και κατέληξε σε συμπεράσματα σχετικά. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και το Συμβούλιο Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων στις 19 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα τα συμπεράσματα. Στα συμπεράσματα αυτά το Συμβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη μέχρι τα τέλη του 2011 να έχουν κάνει τις εθνικές τους στρατηγικές για τη συμπερίληψη των και να βελτιωθούν οι πολιτικές και να ενσωματωθούν και στις υπόλοιπες. στρατηγικές αυτές θα πρέπει πρώτα να καταγραφεί η κατάσταση την οποία βιώνουν ε, οι Ρωμά στα διάφορα κράτη-μέλη. Στα τέσσερα θέματα που σας ανέφερα, παιδεία, στέγη, απασχόληση και υγεία. Και τα κράτη-μέλη στη συνέχεια θα πρέπει μέχρι τέλη του έτους να καθορίσουν τη στρατηγική τους και να εκπονήσουν σχέδια. Επίσης, το Συμβούλιο ζήτησε να χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι με καλύτερο τρόπο. Μετά την έγκριση, λοιπόν, αυτών των συμπερασμάτων, τόνισαν και τα κράτη-μέλη ότι δεσμεύονται να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, σημαίνει προστιθέμενη αξία. Τώρα, μπορεί να με ρωτήσετε τι σημαίνει η δέσμευση των κρατών μελών στην πράξη. Σημαίνει ότι είναι διατεθειμένα να μεταξελιξούν και να αναπτύξουν περαιτέρω τη στρατηγική για τους Ρωμά και μέχρι τα τέλη του έτους να έχουν εγκρίνει ένα πακέτο μέτρων. Μια δέσμη μέτρων υπέρ των Ρωμά και δεσμεύτηκαν, επαναλαμβάνω, τα ε, κράτη-μέλη να συντονίζονται μεταξύ τους την προσπάθεια αυτή και να την εντείνουν. Και προϋπόθεση για να έχουμε αυτά αποτελέσματα είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ε, δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών. Κάτι άλλο που τόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολύ σημαντικό είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εναρμονίσουν και ε, τις νομοθεσίες τους προς την κατεύθυνση αυτή. Ασχολήθηκε στις 12 Απριλίου και ε, το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και όπως σας είπα στις 19 Μαΐου το Συμβούλιο Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας και Αθλητισμού την επομένη στις 20 Μαΐου. Και το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας ε, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου ε, των ε, Ρωμά, των παιδιών δηλαδή, των μαθητών που φεύγουν νωρίτερα από το σχολείο. Στις 23 Μαΐου εγκρίθηκαν και εκεί συμπεράσματα ε, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τα εξετάσει στις 24 Ιουνίου. Ελπίζουμε δε αυτή η στρατηγική να αποφασιστεί και σε στα, στα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο δηλαδή. Θα ακολουθήσει ένα έγγραφο για την κοινωνική ε, ένταξη το Ρωμά. Στο τέλος θα ήθελα να σας πω ότι ε, πρέπει να δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας ζωντανή. Πολλοί από εσά θα αναρωτηθείτε, ωραία, έχουμε μια νέα στρατηγική πλαίσιο, θα λύσει αυτά τα προβλήματα το Ρωμά. Εντάξει, είναι ρητορική ερώτηση. Καταλαβαίνετε ότι η απάντηση θα δοθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτή η στρατηγική βεβαίω είναι ένα πρώτο βήμα, δεν είναι καθόλου πανάκια και σε καμία περίπτωση η λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εκδίδει έκθεση παρακολούθηση ετησίως και θα την παρουσιάζει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Minister. Now... Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Ο πρώτος γύρος για τις πολιτικές ομάδες. Και αν θέλετε μπορούμε να έχουμε και δεύτερο γύρο. Και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβει το λόγο για κάποια σημεία που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση του Υπουργού. Το θέμα της ένταξης των Ρωμά είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Φαντάζομαι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει κάτι να πει. Ελπίζω δηλαδή, ρωτάω. Thank you, Mr. Chairman. Well, I have to start... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για τις άοκνες προσπάθειές της, τη δέσμευσή της ε, για το θέμα αυτό και την υποστήριξή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και να πω ότι αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αποτελούν ορόσημο για το θέμα της ένταξης των Ρωμά. Ε, δεν μιλούμε πια για ένα απλό έγγραφο ή μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα τομέα που εκπίπτει των αρμοδιοτήτων της. Πρόκειται για μια συνεργασία, για ένα κοινό εγχείρημα των τριών θεσμικών οργάνων. Και παρά τις πολλές νομοθετικές προτάσεις, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει κάποια θέματα στα κράτη-μέλη, είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που τα κράτη-μέλη συνένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να επιλύσουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, ήδη ε, είπατε ότι είναι ρητορικό το ερώτημα αν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ή η ανακοίνωση αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα. Όχι βέβαια. Απλώς αποτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα την αρχή μιας χρονοβόρας διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι μας και ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορούμε να αντικρίζουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε, ανέλαβε την υποχρέωση να διεξαγάγει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και να ενημερώσει να ενημερώνει κάθε χρόνο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ευελπιστώ για να μην πω ότι πιστεύω ακράδαντα με τέτοια βεβαιότητα όπως αυτή που βρίσκομαι εδώ σήμερα εδώ, ότι κάθε χρόνο θα έχουμε πρόοδο για να σας αναφέρουμε σε αυτές τις αιτήσεις ενημερώσεις. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες Πρώτα ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ, ο κύριος Δίας Δεβέρα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Υπουργό, τον κύριο Μπάλοκ, για την ε, παρουσίασή του. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία για τις εντυπωσιακές προσπάθειες ό,τι αφορά την ένταξη αυτής της σημαντικότερης μειονότητας που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της μειονότητας των Ρωμά. Και στην Ισπανία έχουμε μια ισχυρή και ιστορική δέσμευση απέναντι στη μειονότητα αυτή, προκειμένου να πετύχουμε όλο και μεγαλύτερα, υψηλότερα ποσοστά κοινωνικής ένταξης. Και μάλιστα έχουμε πολύ... Εγώ είχα και πολύ προσωπικές θετικές εμπειρίες ως δήμαρχος της πόλης μου, στα θέματα αυτής της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Όπως είπατε κι εσείς, όταν μιλούμε για την ένταξη, δεν θα πρέπει να μιλούμε το θέμα της παιδείας, της υγείας, της απασχόλησης και της στέγης. Αυτά τα τέσσερα, αυτοί οι τέσσερις πυλώνες είναι σαν τα τέσσερα πόδια απαραίτητα θεμέλια της ένταξης. Έχω όμως και κάποιες ανησυχίες μετά από κάποια φαινόμενα που παρατήρησα και σε άλλες χώρες Ευρώπης και στη δική μου πατρίδα. Σε αυτό το έγγραφο για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά στην Ευρώπη φαίνεται ότι σημαντικό είναι να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε ε, την συμπερίληψη σε αυτό το δημοτολόγιο. Επίσης, στις απογραφές που γίνονται από τους Δήμους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο σημείο αυτό προκειμένου να προωθήσουμε και το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε και των ε, μελών της κοινότητας Ρωμά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που δεν σχετίζονται μόνο με την κοινωνική ένταξη, αλλά και την εξασφάλιση της συμμετοχής της μειονότητας των Ρωμά στον ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτικό βίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έντσιου από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον ε, Υπουργό Παλούκ για τις ε, υποδείξεις του σε σχέση με την κατάσταση ως προς το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο εκ πρώτης όψεως ίσως δεν φαίνεται τόσο σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι α, αλλά από καιρού καιρών αποδεικνύεται πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα υπό την οπτική γωνία της ένταξης των Ρωμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία διότι κατάφερε να προωθήσει αυτή την στρατηγική πλαίσιο καθώς και την Ευρωπαϊκή Επίτροπη και ιδιαίτερα την Επίτροπο Ρέντιν η οποία μέσω της ανακοίνωσής της ενέταξε σε αυτή τη στρατηγική ένα άλλο σημείο που το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή έτσι ώστε οι κοινότητες των Ρωμά να γίνουν κοινωνοί, διότι όποια άλλη στρατηγική θα παραμείνει νεκρό γράμμα. Γι' αυτό από προσωπικής πλευράς και από πλευράς χριστιανοδημοκρατών θεωρώ ότι σε αυτή τη στρατηγική αυτή η στρατηγική μάλλον θα πρέπει να μεταφερθεί in situ, δηλαδή να υπάρχει ένας διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινότητας, Ρωμά και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Χωρίς, Χωρίς αυτό το τρίο, καμία στρατηγική δεν θα μπορέσει να επιτύχει για αυτή την εθνοτική μειονότητα. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί από την πείρα μου, τουλάχιστον στη Ρουμανία από όπου προέρχομαι και όπου έχουμε πολλές ε, κοινότητες Ρωμά, όλες οι εθνικές στρατηγικές δεν είχαν ε, αυτά αποτελέσματα μέχρι τούδε, διότι αυτές οι στρατηγικές ε, δημιουργήθηκαν στα γραφεία από υψηλούς αξιωματούχους με μεγάλη προετοιμασία, χωρίς όμως να έχουν ε, πρακτική έμπρακτα πείρα οι εμπειρίες. Και εγώ ήμουν αντιδήμαρχος του Βουκουρεστίου. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα Ρωμά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι και η μόνη η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτής της κοινότητας και να αναγνωρίζουν έμπρακτα τις ανάγκες τους, την ανάγκη αυτής της μεγάλης κοινότητας. Αυτή είναι λοιπόν η, αυτή θα πρέπει να είναι οι άξονες δηλαδή εκπαίδευση, στεγαστικό, υγεία, υποδομές. Αυτοί είναι τέσσερις πυλώνες, αν θέλετε, στους οποίους θα πρέπει να βασιστούμε για να προωθήσουμε τις δραστηριότητες μας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινότητα των Ρωμά δεν συμμετείχε έμπρακτα σε καμία από αυτές τις στρατηγικές. Δηλαδή δεν ήταν κοινωνή η Ρωμά. Και δυστυχώς όλες αυτές οι στρατηγικές πλαίσιο δεν λαμβάνουν υπόψη ότι αυτή η εθνότητα έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι νομάδες, έχουν υψηλή κινητικότητα. Δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο. Πρόκειται για μία εθνότητα νομάδων και γι' αυτό η στρατηγική αυτή θα έπρεπε να λάβει υπόψη αυτό το νομαδικό χαρακτήρα και την υψηλή κινητικότητα των ε, Ρωμά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών. Για παράδειγμα, συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ρουμανίας έτσι ώστε από κοινού να δημιουργήσουν κοινέ υποδομές. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, αφορά και άλλες χώρες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν από κοινού προγράμματα για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, είτε θέλουν να εγκατασταθούν στη Γαλλία είτε στη Ρουμανία. Χρειάζεται συνεργασία των κρατών μελών. Ε, διαφορετικά δεν θα στεφθεί από επιτυχία η στρατηγική μας. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι στη Ρουμανία δεν μπορώ να μιλήσω για την Ουγγαρία, για άλλες χώρες. Εάν η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινότητα των Ρωμά και η κοινωνία των πολιτών δεν θα συνεργαστούν, αν δεν υπάρχει συνεργασία αυτή τη τριάδας δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί καμία στρατηγική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλτέρα από τους Φιλελεύθερους. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του και την Ουγγρική Προεδρία μετά το εξάμενο που ήταν επιτυχές και δίνει κάθε λόγο ικανοποίησης στην Προεδρία για τη στρατηγική των Ρωμά. Νομίζω ότι όποιο και αν ασκεί την Προεδρία, το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ούτε σε ένα εξάμεινο, ούτε καν σε μία εξαετία. Πρόκειται για μία μακρόπνοη στρατηγική αυτή που εγκαινιάζουμε τώρα και όλες οι μελλοντικέ προεδρίες έχουν κάτι να πούν για το θέμα. Για μας τους φιλελεύθερους είναι σημαντικό να μην ε, ασχοληθούμε μόνο με το οικονομικό σκέλος, γιατί θα είναι χρήσιμα φυσικά τα κονδύλια, αλλά το πιο σημαντικό είναι να προσαρμόσουμε και να εφαρμόσουμε τις ε, κατάλληλες νομοθεσίες. Δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα συμπεριφοράς και να δώσουμε την αίσθηση να πείσουμε τους Ρωμά ότι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, ότι έχουν ίσες ευκαιρίες και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό δεν μπορεί να επιληθεί με κανένα ποσό χρηματικό αφορά τις τοπικές κυβερνήσεις και είναι δική τους ευθύνη. Νομίζω ήταν σωστή και η στάση της κυρίας Ρέντινγκ, της Επιτρόπου Ρέντινγκ, ευθύς εξ αρχής και είναι λογικό να αισθάνεται και πάλι η περήφανη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, είναι πρόημο από τώρα να θριαμβολογούμε. Θα δούμε σε μία δεκαετία αν όντω έχουμε λόγους να είμαστε υπερήφανοι για αυτή την πολιτική. Τότε θα κριθούμε. Πάντως καλό είναι να ξεκινήσουμε σε αυτή την πορεία που εγκαινιάσαμε και να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία που εγκαινιάσαμε. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, η κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι για την αισιοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την έκβαση αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά είναι νωρίς ακόμη να είμαστε αισιοδοξοί. Θα το δούμε αργότερα, γιατί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα διακριτικής μεταχείρισης βάρος των Ρωμά χρόνια ολόκληρα, για να μην πω δεκαετίες ολόκληρε. Και δεν μας έλειψαν ούτε διακηρύξει, ούτε διασκέψεις κορυφής για το θέμα αυτό, ούτε κονδύλια. Πολλά λόγια, αλλά ελάχιστες αλλαγές. Και σε πολλές χώρες μέλη οι Ρωμά είναι θύματα διακρίσεων, περιθωριοποιούνται συστηματικά, δεν έχουν πρόσβαση και μάλιστα είχαμε και τις ε, πρόσφατες απελάσεις από τη Γαλλία. Πολλά είναι τα αρνητικά παραδείγματα. Πάντως είναι καλό ότι αποτέλεσε το θέμα αυτό προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας. Αυτό αν μη τι άλλο είναι θετικό. Είναι σημαντικό όμως ταυτόχρονα μια Προεδρία να δώσει και ένα παράδειγμα προς μίμηση, να γίνει ένα υπόδειγμα για τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυση των προβλημάτων. Περιμέναμε πολύ περισσότερα από την Ουγγρική Προεδρία. Να σταματήσουν αυτά τα συλλαλητήρια των ναζιστών ε, ε, ή να αποστέλλονται οι Ρωμά για θερινές διακοπές εντός εισαγωγικών για τις οποίες δεν έχουν ιδέα. Πολλά από αυτά που έγιναν στην Ουγγαρία φυσικά δεν φταίτε εσείς. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αντισταθεί, να αντιταχθεί, να περιορίσει αυτές τις ομάδες, να, είναι, να δείξει πυγμή στην προσπάθεια καταπολέμησης τους. Και από αυτή την άποψη θα μπορούσε να είναι πιο αποφασιστική στη στάση της Ουγγρική κυβέρνηση. Η Ουγγρική κυβέρνηση. Ε, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, πολύ συχνά το Συμβούλιο ξεχνά ότι η βάση της ένταξης είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη μυσαλλοδοξία εις βάρος των τσιγκάνων, των Ρωμά, να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το θέμα της στέγασης, γιατί ακόμη και αν εσείς νοικιάζετε το σπίτι σας σε μια οικογένεια Ρωμά που στη συνέχεια θα υποστούν τις λιδωρίες των γειτόνων, δεν έχει νόημα δεν είναι μόνο το θέμα η σωστή πολιτική, είναι να καταπολεμούμε τη διάκριση όπου και αν εμφανίζονται και από τους ε, ναζιστές και στο δρόμο, οπουδήποτε και στα θεσμικά όργανα. Από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και πιο συγκεκριμένοι, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε άμεσα και αυτά αποτελέσματα. Νομοθεσία έχουμε ήδη, δεν χρειάζομαστε τίποτα καινούριο, απλώς θα πρέπει να την εφαρμόζουμε. Και νομίζω ότι εκεί είναι που υπάρχουν κενά. Εν πάση περιπτώσει, μια και θέλουμε να δείξουμε αισιόδοξη και εγώ ευελπιστώ ότι η πρόοδος από εδώ και πέρα θα είναι ταχύτερη. Αλλά μέχρι στιγμής ήταν προαιρετική αυτή η διακήρυξη των κρατών μελών. Δεν προβλέπονται ούτε πιθανότητες επιβολής κυρώσεων, τίποτα. Ελπίζω τουλάχιστον στην έκθεση να μην λέμε όλα είναι ρόδινα και αγγελικά πλασμένα, να επισημαίνουμε τα λάθη, τα κενά, τις αδυναμίες και τα σφάλματα των κρατών μελών, γιατί αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενό σωστού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστ. Διαπιστώνω ότι ο χρόνος που έχουμε προβλέψει για τη συζήτηση με τον ε, Ούγγρο Υπουργό είναι μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Θα έλεγα να συγκεντρώσουμε όλες τις ερωτήσεις και μετά να δώσει απάντηση ο Υπουργό. Δεν θα έχουμε δύο γύρους. Θα δώσω το λόγο στον, στην κυρία Ένστ πρώτα και μετά στον κύριο Μπρόνς. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό. Καταρχάς γνωρίζω ότι ήταν πάρα πολλές οι πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Κάνατε πολλές προσπάθειες να προωθήσετε τα θέματα αυτά. Βέβαια, σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα δεν μπορεί κανείς να επιτύχει τα πάντα. Σωστό είναι αυτό. Και χαίρομαι που μιλήσετε και ειλικρινά ε, για αυτό το πρόβλημα της στρατηγικής πλαισίου. Και θα πρέπει και εδώ να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς και εμείς και να πούμε, όπως είπατε και εσείς, ότι δεν αρκεί, ότι δεν είναι ούτε πανάκια ούτε λύνει τα προβλήματα. θα πρέπει να κινηθούν τώρα τα κράτη-μέλη. Είναι καλή στρατηγική ε, πλαίσιο και ε, βασίζεται σε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι Λίβια. Τώρα λοιπόν καλούνται τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν αυτά και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τόσο μεγάλες οι προσδοκίες και οι ελπίδες που έχουν αποθέσει η κοινότητα το Ρωμά πλέον ε, στα χέρια μας, ότι θα αλλάξει κάτι, ότι θα γίνουν πραγματικές αλλαγές και μπορούν να γίνουν και θα επέλθουν έτσι κι αλλιώς και θα πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στα κράτη-μέλη γιατί αν αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη, για χρόνια ολόκληρα θα μείνουμε πίσω και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, ε, μιλήσατε για αιτήσια έκθεση παρακολούθηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ δεν θέλω να έχουμε μια έκθεση μόνο, δεν μου αρκεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εδώ στο Κοινοβούλιο δηλαδή, θα πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε τι θα γίνει από συγκεκριμένα βήματα μετά τις εκθέσεις αυτές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μπορεί να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται τελείως διαφορετική προσέγγιση πέρα από τη στρατηγική πλαίσιο και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε προβλέψει. Σε ευρωπαϊκό επαναλαμβάνω επίπεδο. Και να είμαστε και ειλικρινεί και σαφείς και να τα λέμε και στα κράτη-μέλη με το όνομά τους τα πράγματα. Μετά από κάθε έκθεση προόδου, παρακολούθησης, πώς θα λέγεται, να δεσμευτούμε να κάνουμε κάτι, να δίνουμε συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτον, η συμπερίληψη και η ένταξη των Ρωμάτων, τον ίδιο το είπε και ο κύριος Έντσιου. Δεν πρόκειται να κινηθεί τίποτα εάν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τους Ρωμά να ενδιαφερθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για θέματα που τους αφορούν. Μήπως χρειάζεται και αναδιάρθρωση εδώ, υποδομές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών όμως. Να αναλαμβάνουν τους ευθύνες του ήδη να συμμετέχουν. Και εγώ θα ήθελα και ένα ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο Ρωμά και να κάνουμε κάθε φορά μια καταγραφή. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, πώς έχουμε προχωρήσει στα κράτη-μέλη, πού φτάσαμε, τι απομένει. Ένας ετήσιος απολογισμός και να το πιέσουμε. Όχι να περιμένουμε κάθε χρόνο πότε θα μας έρθει η ωραία έκθεση που θα μας τα λέει ε, όμορφα. Να τονίσουμε ότι χρειάζεται πίεση, να την αυξήσουμε την πίεση και να κάνουμε κάτι. Το τελευταίο. Καταπολέμηση των διακρίσεων. Εντάξει, αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα. Η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν είναι το αντικείμενο βέβαια της στρατηγικής πλαισίου αποκλειστικά. Ε, ίσως χρειάζεται και μια εκθέση πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζονται ειδικά προγράμματα για την άρση των ε, διακρίσεων ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό βοηθάει καλύτερα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ξέρω ότι το χρήμα δεν είναι το παν, υπάρχουν και άλλα ε, βήματα που μπορούν να γίνουν και πάρα πολύ αξιόλογα αυτά. Mr. Ο κύριος Μπρόνς έχει Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί που μιλάνε υπέρ των μέτρων είναι πολύ γενναιόδοροι άνθρωποι, αλλά η προσέγγιση τους ε, είναι κάπως αυταρχική και ίσως δεν λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο χαρακτήρα αυτών το μέτρο. Δηλαδή, ε, δεν μιλάμε για το... Ε, δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν άψυχα ε, όντα, τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να αλλάξουν τον κόσμο τους ε, μόνοι τους. Αυτό ε, έχει σχέση με το γεγονός ότι οι άνθρωποι γεννιούνται τα μπουλαράζα και μετά ε, αποκτούν όλα δηλαδή τα άλλα είναι επίκτητα. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, ο πολιτισμός είναι απότοκο μίας γενικότερης προσέγγισης των ανθρώπων. Οι Ρωμά έχουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά αυτό το σχετίζεται με τις δικές τους προσπάθειες και όχι ε, και δεν αφορά το τι έρχεται από τα πάνω. Η κοινότητα, η Βρετανική κοινότητα των ε, Ρωμά είναι ξεχωριστή και υπάρχει μία γενεαλογική εξέλιξη αυτής της κοινότητας. Δυστυχώς όμως μπορούμε να πούμε ότι η κοινότητα ε, Ρωμά εμπλέκεται σε εγκληματικές ε, δραστηριότητες πολλές φορές. Και ρώτησα ένα χρόνο πριν τον εκπρόσωπο της Europol στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ κατά πόσο υπάρχει πραγματικά αυτή η εμπλοκή και κατά πόσο υπάρχει και εμπορία ανθρώπων από αυτή την κοινότητα. Ε, μου ελέγχθη, η απάντηση μάλλον ήταν καταφερτική και είπα ότι το πρόβλημα και αυτή του, η πτυχή του προβλήματος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρόεδρος, εάν κανένας άλλος δεν θέλει να λάβει το λόγο, θα ακούσουμε τώρα την απάντηση στα ερωτήματα αυτά από τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για τη δραστηριότητά τους. Eh, έχει μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη σημασία να ακούμε και όχι να μιλάμε. Γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος στις απαντήσεις μου. Θα ήθελα να ε, ε, πω στον Ισπανό βουλευτή ότι γνωρίζω ότι στην Ισπανία υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες και αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετοχή της κοινότητας. Βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι πρόκριμα δηλαδή. Αυτοί οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο ληξιαρχείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε τι θα κάνουμε και στη Ρουμανία με τους Ρωμά. Κανένας δεν μπορεί να τους σταματήσει ως προς την κινητικότητα και γι' αυτό θα πρέπει να ε, τους βοηθήσουμε. Αλλά πρόκριμα γι' αυτό είναι να έχουν εγγραφεί στο ληξιαρχείο. Ο κύριος Έντσιου μίλησε για τις ε, τοπικές αρχές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την ομαδική εργασία. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι έγινε μια δημοσκόπηση στην Ουγγαρία πρόσφατα από όπου ανακύπτει ότι οι Ρωμά έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις τοπικές αρχές. Δηλαδή στις τοπικές αρχές, στον δήμαρχο, στα σχολεία, στο διευθυντή του σχολείου, στον ε, γιατρό, στον οικογενειακό γιατρό και ούτω καθεξής. Πολύ περισσότερο από ό,τι εμπιστεύονται τις εθνικές αρχές. Σε σχέση με την κινητικότητα θα ήθελα να πω ότι Ίσως η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, όμως στην Ουγγαρία εδώ και τρεις γενές οι Ρωμά έχουν εγκατασταθεί και δεν παρουσιάζουν αυτό το νομαδικό χαρακτήρα. Αλλά βεβαίως μπορούμε να συνεργαστούμε και με άλλες χώρες όπως η Γαλλία σε περιπτώσεις κινητικότητας. Ε, κύριε Μούλτερ, η βασική οργάνωση η οποία ασχολείται ε, με τους Ρωμά στην Ουγγαρία φέρει το όνομα The Lungodrom. Lungodrom σημαίνει ε, ένας μακρύς δρόμος που απαρτίζεται από πολλά μικρά βήματα. Και αυτή η οργάνωση ασχολείται επισταμένως με τους Ρωμά. Η κυρία Κέλλερ μίλησε για τα μέτρα τα οποία εγκρίνονται ή οφείλουν να εγκριθούν. Οι Ρωμά θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζονται όχι πατερναλιστικά, αλλά σαν έμψυχα όντα, σαν αυτοτελείς οντότητες οι οποίες έχουν ε, λόγο και έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες ε, όπου μπορούν να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους οι Ρωμά και τους ε, εκλέγουν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα σε εθνικό επίπεδο μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντα της κοινότητάς τους. Και ο Πρωθυπουργό έφτασε σε μια συμφωνία με, τον, ε, με τους επικεφαλείς των Ρωμά στις διάφορες κοινότητες Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα, σύστημα, ένα εθνικό σύστημα λήψης αποφάσεων όπου αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες. Προσπαθούμε λοιπόν να λάβουμε αποφάσεις μετά από διαβουλεύσεις και σε τέσσερα χρόνια έχουμε υποσχεθεί να εντάξουμε στην αγορά εργασίας 100.000 Ρωμά και σε τέσσερα χρόνια θα έχουμε 5.000 νέους ρωμαθητητές που θα φοιτούν στα πανεπιστήμια μας. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να μεταφερθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε επαρκώς αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχει νόημα να προβάλλουμε ε, διεθνείς στρατηγικές ή εθνικές στρατηγικές. Ως προς την υπόδειξη του μέλους που μίλησε για την ε, καταπολέμηση των διακρίσεων, υπάρχουν ε, μη κυβερνητικέ οι οποίες επέκναν την Επιτροπή για την ανακοίνωσή της. Αν δείτε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, βλέπετε ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα χάσματα που υπάρχουν και στα συμπεράσματα βλέπουμε ότι το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να ε, εποπτεύσει αυστηρά την εφαρμογή της οδηγίας κατά των διακρίσεων και δυνάμει της οδηγίας αυτής υπάρχουν αποδοτικά μέσα για την καταπολέμηση των διακρίσεων ανάλογα με την εθνοτική προέλευση. Αυτό αποτελεί απαράβατο όρο για την ένταξη και των Ρωμά. Και στα έγγραφα αυτά σε σχέση με την, με την εκπαίδευση και την ένταξη των Ρωμά ε, μιλήσαμε για τα επιμέρους ζητήματα που μας απασχολούν, δηλαδή την εκπαίδευση, τον τομέα της υγείας και ούτω καθεξής. Επίσης μας απασχολεί και το θέμα των θέσεων εργασίας, της απασχόλησης. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να ειδωθούν από κοινού και όχι να θέσουμε τη μία διάσταση κατά της άλλης. Τώρα, ως προς τις νεοναζιστικές οργανώσεις στην Ουγγαρία, έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο ανακύπτει παντού στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ουγγαρία. Δυστυχώς, οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά ανάλογα με τις περιστάσεις υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλουν να στυλιτεύσουν αυτή την κατάσταση και να, και να καταπολεμήσουν τις ε, ε, μειονότητες. Αυτές οι προκλήσεις άρχισαν το ε, Μάρτιο στην πόλη Γκιονγκεσπάτοκ και στις 2 Μαΐου στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο εγκρίναμε έναν νέο νόμο για την ε, καταπολέμηση, την δίωξη αυτών των αδικημάτων, έτσι ώστε να μην εκφοβίζεται καμία μειονότητα και να καταπολεμήσουμε και αυτή την απαράδεκτη στάση των νεοναζιστών. Εγώ για τέσσερα χρόνια ασχολήθηκα με αυτό το θέμα στην ε, Ουγγαρία θα πρέπει να εξευρεθεί μια λύση έτσι ώστε να μην υπάρχει, ε, να μην υπάρχει δυνατότητα, η ελεύθερη δυνατότητα του εκφράζεστε. Πρόκειται για παράβατα δικαιώματα. Επίσης, το θέμα της απασχόλησης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διότι γνωρίζετε ότι από πλευράς αστυνομίας καταβλήθηκε μία προσπάθεια, δηλαδή έγιναν συλλήψεις, αλλά τελικά οι πολίτες αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως ήταν ιδιαίτερα δραστήριο τις τελευταίες εβδομάδες. Βρέθηκε σε πολλές πόλεις και οι Ρωμά εξέφρασαν την θέλησή τους να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι η εποπτεία είναι πολύ σημαντική. Εάν τεθεί σε εφαρμογή σωστά αυτή η εποπτεία, τότε η στρατηγική μας θα στεφτεί από επιτυχία. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται μόνο λεκτικές επικρίσεις, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε τους μηχανισμούς που θα ε, έχουν σαν συνέπεια και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων. Αυτή η πρωτοβουλία της Ουγγρικής Προεδρίας θα πρέπει να οδηγήσει σε μία πλατφόρμα η οποία θα λάβει θεσμικό χαρακτήρα. Στη Βουδαπέστη είχαμε 400 εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της κοινότητας των Ρωμά. Κατά τη γνώμη μου αυτό το πλαίσιο μπορεί να διευρυνθεί έτσι ώστε κάθε έξι μήνες να υπάρχει δυνατότητα ε, διοργάνωσης διασκέψεων και σεμιναρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Μπρόν στη συνέχεια μίλησε για τον κίνδυνο αυτό της επιβολής ε, μέτρων εκ των άνω. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη τις ίδιες, την ίδια τη μορφή οργάνωσης των ορμά. Κατά την άποψή μου, έχει μεγάλη σημασία να δούμε και τις εργασίες του Συμβουλίου, διότι μας ενδιαφέρει η καταπολέμηση του εγκλήματος και της εμπορίας προσώπων. Και έτσι το θέμα προσλαμβάνει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο κοινός μας αγώνας κατά, της, ε, κατά του εγκλήματος και της δουλείας καθώς και της εμπορίας προσώπων. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες προωθούν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες μεταξύ αυτών των θυμάτων οι Ρωμά αποτελούν πολύ υψηλό ποσοστό. Πρόκειται δηλαδή για μια ευάλωτη κατηγορία. Φέρουμε κοινή ευθύνη λοιπόν για την προστασία τους. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας, για την αποκοινού εργασία Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούμε επικρίσεις για ένα θέμα που μας απασχολεί και στο οποίο, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Χρειαζόμαστε συμμάχους και όχι επικριτές και για την ε, ένταξη των Ρωμά και για την καθημερινή μας εργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχω την υποστήριξή σας έτσι ώστε κατά την προσεχή Προεδρία και τις ε, προεδρίες ε, στη συνέχεια, το θέμα αυτό θα αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής διότι η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας των Ρωμά είναι κάτι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν βοηθήσουμε τις ευάλωτες αυτές κατηγορίες, τότε ε, τίθεται ένα αμφιβόλο η γενικότερη μας πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την ειλικρίνειά σας, την ε, προθυμία σας για συνεργασία, την ε, αγαστή συνεργασία που είχατε με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Διαπιστώσατε ότι και εμείς ε, δεχθήκαμε και επιδοκιμάσαμε τις προτάσεις σας για την κοινωνική ένταξη, για τα ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ένταξη των Ρωμά στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες Ευρώπης που έχουν σημαντική παρουσία αυτής της μειονότητας. Είναι σημαντικά όλα αυτά και χθες είπαμε στους υπουργούς ε, Πίντερ και Ναβράτσιτς Υπουργού Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων. Καλή τύχη. Το ίδιο λέμε και σε εσά. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία στην τελική φάση της Ουγγρική Προεδρία και καλή τύχη και στα πλαίσια του τρίου στη συνεργασία με την Πολωνική Προεδρία για να συνεχίσετε αυτή την ε, πολιτική που ξεκινήσατε. Σα ευχαριστούμε. And now... Περάμε τώρα στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης. Έχουμε εδώ ένα θέμα που εμπίπτει σε κοινή αρμοδιότητα και τη Επιτροπή Απασχόληση, για ορισμένα τουλάχιστον σημεία, για ορισμένε πτυχές. Ο δικός μας ηγετή είναι ο κύριος Γιακολίνο. Θα εξετάσουμε το σχέδιο εκθεσή του και θα ορίσουμε και την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Το θέμα αυτό των επιχειρησιακών αποσπάσεων ακολουθεί μετά από ακρόαση που είχαμε οργανώσει τον Απρίλιο, σε αρχές Απριλίου και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις θέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουγγρικής Προεδρίας, αλλά και την ε, θέση της κυρίας Γεκονσάρη, που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης. Πρώτο όμως, το λόγο θα έχει ο δικός μας ηγετής, ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ πολύ καλά υπενθυμίσατε ότι πρόσφατα διοργανώθηκε μία ακρόαση από τη Γραμματεία όπου συζητήσαμε το θέμα αυτό της ε, προστασίας των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια των ενδεχομένων αποσπάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει αυτό το θέμα και μέσα στα πλαίσια του ενδοκοινοβουλευτικού διαλόγου. Πρόκειται για ένα πακέτο το οποίο παρουσίασε η Επίτροπος η κυρία Μάλστρεμ για τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να ορίσουμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν την μπλε κάρτα και άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν σε συνέχεια, δηλαδή ως προς τους εποχικούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι συμβαίνει ιδιαίτερα στη Μεσόγειο έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την υποδοχή και την ένταξη δυναμικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές απαιτήσει της αγοράς. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Το είδαμε με την κυρία Γιάν Κονσάρη και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την αρρωγή της. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης προβλέπει αυτή την παρέμβαση η οποία ε, αρθρώνεται με βάση ένα έγγραφο όπου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε υπόψη το άρθρο 50. Με τον πρόεδρο φτάσαμε σε ένα συμβασμό προς το άρθρο 3 καταρχήν έτσι ώστε να υπάρχει ορισμός των ε, κατηγοριών εργαζομένων είτε πρόκειται για διευθυντικά ε, στελέχη, είτε πρόκειται για εργαζόμενους κατωτέρων βαθμίδων. Εγώ υπέβαλα ορισμένες ε, τροπολογίες έτσι ώστε να γίνει πιο εύληπτο ένα έγγραφο το οποίο έχει ολένα και μεγαλύτερη πολιτική σημασία. Μας ενδιαφέρει η προστιθέμενη αξία κάθε επιχείρησης η οποία χρειάζεται έμψυχο υλικό και το οποίο δεν μπορεί να αποκτήσει διαφορετικά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι σημαίνει διευθυντικό στέλεχος, τι σημαίνει εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να έχουμε ένα ομοιόμορφο πλαίσιο και θεωρήσαμε ότι τη στιγμή που το θέμα της εμπιστοσύνης, αμοιβέ εμπιστοσύνης προσλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, το κριτήριο αυτό δεν μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο μέσα σε ένα τέτοιο έγγραφο. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς ορίζεται το πλαίσιο αυτό της ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης, ακόμα και σε τρίτες χώρες θεωρήσαμε ότι το διευθυντικό προσωπικό θα πρέπει να προσλαμβάνεται με βάση μετρήσιμα ε, στοιχεία και να δούμε και ποια είναι η πείρα αυτού του προσωπικού. έχουμε λάβει υπόψη το κοινοτικό προτιμησιακό καθεστώς και μιλάμε και για την οικογενειακή επανένωση, δηλαδή ε, ε, αν μιλάμε για απόσπαση σε τρίτες χώρες. Επίσης, αυτό μας ενδιαφέρει είναι η προγενέστερη απασχόληση στην επιχείρηση που θα ορίζει και την απόσπαση. Δηλαδή, η απασχόληση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξαμηνιαία για να μην γίνουν καταχρήσεις. Μας ε, ενδιαφέρει και η εποπτεία και ο έλεγχος έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός και η άδεια παραμονής θα πρέπει να οριστεί με ένα ενιαίο έγγραφο μαζί με, ε, με τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα για την απασχόληση ως προς του... τις επιχειρήσεις ή του ομίλους επιχειρήσεων θα πρέπει να δούμε τι ορίζει το άρθρο 16. Το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει αποφανθεί. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και με τις τροπολογίες και θα σας ε, παρουσιάσω ενδεχομένως και άλλες. Πέρα από την ε, απόσπαση, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς αυτοί οι εργαζόμενοι με πολύ ψηλά ε, προσόντα μπορούν να αποσπαστούν για μια περίοδο η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τροπολογίες έτσι ώστε να διαμορφώσουν καλύτερα το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έχει ήδη γίνει μια αξιολόγηση και μελέτη επιπτώσεων και αναμένοντας ε, τις τροπολογίες των ε, μελών, των σκιωδών και ούτω καθεξής, πιστεύουμε ότι θα διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο. Το έγγραφο αυτό θέλουμε να είναι εύληπτο και να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Ξέρω ότι θα επανέλθει επί του θέματος στο Συμβούλιο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών. Τις επόμενες εβδομάδες θα επανέλθουμε επί του θέματος. Θα σταματήσω εδώ, λοιπόν, έτσι ώστε να ακούσω και τους άλλους και ελπίζω, αφού ακούσουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε νέα στοιχεία ή συμπληρωματικά στοιχεία πλαισίωσης. Αυτό το θέμα ε, αφορά και τους εποχικούς, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά δεν είναι τόσο ε, περίπλοκο για τους εποχικούς. Γι' αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, υπάρχουν ανώτατα διευθυντικά, ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τα οποία να μπορούν να αποσπαστούν με ευκολία. Αυτά, αυτό είναι το σκεπτικό μου, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των εργασιών. Τώρα προτείνω να ακούσουμε την Επιτροπή, από την Επιτροπή και την Προεδρία. Για ε, και την ε, εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης, κυρία Γιακονσάρη. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση αυτής της ε, ακρόαση. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη για να προχωρήσουμε στις εργασίες μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή του κύριο Γιακολίνο. Τώρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο ε, επί της προτάσεως αυτής. Όπως είπε και ο κύριος Γιακολίνο, είναι συνολικό πακέτο συλλογικής στρατηγικής για την πολιτική μετανάστευση και πιστεύω και ελπίζω να εγκριθεί σύντομα και η πρόταση αυτή και η πρόταση για τους εποχικούς εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά τις ενδοεπιχειρησιακές αυτό έχει και ένα θέμα και ρόλο να παίξει για τη στρατηγική του 2020. Ε, και η τεχνολογία της, ε, πληροφορίας, της πληροφορικής θα αναπτύξει και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και τεχνολογίας. Ε, έχουν γίνει κάποιες τροπολογίες στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διευκρινίσουν κάποια στοιχεία και να βελτιώσουν το κείμενο για να είναι αυτό το σύστημα ελκυστικό και να καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις. Ενισχύονται από τις τροπολογίες λοιπόν κάποια σημεία του κειμένου. Επίσης, Δεν είναι γαλάζια κάρτα. Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται εντό του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων δεν είναι για μόνιμη εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες εβδομάδες και θα δούμε και ε, ποια τελικά θα είναι η μορφή του ορισμού Χρειάζεται να δοθεί μεγάλη προσοχή για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βασιστεί και σε εφισταμένους ε, ε, διορισμούς. Δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι εργαζόμενοι, είναι συγκεκριμένοι ε, άνθρωποι που μετακινούνται στο εσωτερικό ενός ομίλου επιχειρήσεων, είναι στελέχοι και σημαντικά που έχουν μεγάλη επαγγελματική πείρα και μετακινούνται. Δεν είναι τυχαία εργαζόμενοι. Αυτό που θέλαμε είναι αφενός να μην είναι πάρα πολύ περιοριστικό το πεδίο εφαρμογή, αλλά να είναι σαφείς οι ορισμοί όπως σας είπα και ή δυνατόν να βασιστούμε σε ορισμούς που ήδη υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλα σημεία. Η κινητικότητα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζετε ότι είναι πολύ σημαντική ε, είχαμε και άλλες μορφές με τους ε, ερευνητές, με την καλάζια κάρτα, αλλά εδώ για πρώτη φορά συζητούμε αυτό το θέμα, γι' αυτό χρειάζονται διευκρινήσεις και ορισμοί. Στους 12 μήνες προηγούμενης απασχόλησης που έχουμε επιλέξει, στην πρότασή μας ήταν για να αποφύγουμε καταχρήσεις ακριβώς. Αλλά είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Θα περιστώ σε αυτά τα σχόλια προς το παρόν, αλλά βεβαίω δεν είναι χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις αν έχετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Από την Προεδρία, η κυρία Βαλάση. Να σας καλημερίσω και εγώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος της ε, Ουγγρικής Προεδρίας για τη συζήτηση του Απριλίου, η οποία συνεισέφερε καθοριστικά για την πρόθεση αυτού του σχεδίου οδηγίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο για την ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης και πιστεύουμε ότι με αυτό το σχέδιο έκθεσης θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία τάχιστη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η Προεδρία πιστεύει ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική για την νόμιμη μετανάστευση και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εντάχει να σας πω πώς έχει η κατάσταση στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και θα ήθελα να απαντήσω στα επιμέρους σημεία. Όπως είπε ο κύριος Γιακολίνο, είχαμε έξι συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ε, εξαμηνιές προεδρίας και αυτό καταδεικνύει ότι το ζήτημα είναι ύψης της σημασίας για μας, ότι δηλαδή θέλουμε να ε, ασχοληθούμε και να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το σχέδιο οδηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε και στο θέμα της ε, κινητικότητας, ε, διότι το θέμα αυτό μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Το θέμα της ε, Κομισιόν αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του τύπου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών διότι αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε μία αποτελεσματική διαδικασία για την κινητικότητα. Τα στοιχεία αυτά δεν είχαν οριστεί επαρκώς και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή. Προσπαθήσαμε λοιπόν Λοιπόν να βρούμε μια νέα διατύπωση σε σχέση με τη διαδικασία κινητικότητας που να διαφέρει από, το, από τη συλλογιστική της Κομισιόν. Βρήκαμε λοιπόν ένα, ε, νέα ένα, νέο πλαίσιο για την ε, κινητικότητα μέσω και μακροπρόθεσμα. βασιστήκαμε στην ε, οδηγία για το ερευνητικό προσωπικό, ενώ για την κινητικότητα μακροπρόθεσμα βασιστήκαμε στην οδηγία για τις μπλε κάρτες, για τις άδειες εργασίας δηλαδή. Και όπως είπε και ο κύριος Γιακολίνο θα ανακύψουν τροπολογίες επί του θέματος που ελπίζω να οδηγήσουν στην προσέγγιση το, της θέσης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ως προς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, Στις συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας του Συμβουλίου φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να ορίσουμε καλύτερα τις ενδοεπιχειρησιακές αποσπάσεις. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Γιακολίνο ότι θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα το πλαίσιο, να βρούμε καλύτερους και ενιαίους ορισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει μία ενιαία συλλογιστική βάση, η οποία να μπορέσει να εφαρμοστεί εύκολα και αυτό που έχει σημασία είναι να μην υπάρχει περιθώριο διασταλτικής ερμηνείας των άρθρων. Και όσον αφορά τους ασκούμενους, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι περιθώρια υποδοχής υπάρχουν για αυτή την κατηγορία. Αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και οπωσδήποτε θα επιβληθεί μία ελάχιστη ποσόστοση. Ως προς τις συνθήκες υποδοχής, όπως είπε και ο κύριος Γιακολίνο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η περίοδος αναφοράς, η οποία θα πρέπει να μειωθεί από 12 σε 6 μήνες. Η ελάχιστη περίοδος απασχόλησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να βρούμε πιο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης και απόσπασης. Πέρα από αυτό, Το σχέδιο έκθεσης ασχολείται με τις συγκεκριμένες συνθήκες απασχόλησης μέσα στα πλαίσια της ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης. Κατά τη διάρκεια της ε, απόσπασης, ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε και την απασχόληση σε τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν και εντός των κρατών μελών. Όσον αφορά τη την απόσυρση, μάλλον τη μη ανανέωση αυτών των αδειών εργασίας, της μπλε κάρτας δηλαδή, αυτό που έχει σημασία είναι να ορίσουμε καλύτερα το πλαίσιο έτσι ώστε να μην υπάρξουν καταχρήσεις για το μέλλον. Και θα πρέπει να βελτιώσουμε και τις διαδικασίες ανανέωσης. Γι' αυτό χρειάζεται στην οδηγία μέσα σε μία παράγραφο και μόνο να αναφερθούμε σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να έχουμε μία απλουστευμένη διαδικασία για τα κράτη-μέλη που να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αφορά και την ε, απόσπαση μέσα στην ίδια επιχείρηση και την οικογενειακή επανένωση. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο τις, ε, ε, τους ε, πολίτες από τρίτες χώρες, αλλά και τις συνθήκες υποδοχής αυτών των εργαζομένων. Και αυτό θα πρέπει να γίνει εντάχει, μέσα σε 30 μέρες. Επίσης, το Συμβούλιο φτάνουμε σε ένα συμβασμό παρόμοιο με αυτόν στο οποίο φτάσατε εσείς μέσα στα πλαίσια ενός συνενωτικού εγγράφου. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τους φορείς υποδοχής, αλλά και τις πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και για, το, και για το, τη συνέχεια της εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο και ελπίζω να μπορέσουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρας αυτή την εργασία. Ελπίζω αυτή η έκθεση να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για την επόμενη Προεδρία, για την Πολωνική Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ε, εργασία. Βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιακονσάρη, Κονσάρη, εισηγείται στην Επιτροπή Απασχόληση. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιακολίνο ε, πάρα πολύ γόνιμη και χρήσιμη συνεργασία μας. Επανελειμμένα ακούσαμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία εντάσσονται σε ένα πακέτο για τη μετανάστευση. Ωραία, σωστό είναι αυτό. Αλλά τι διαστάσεις έχει προσλάβει, τι όγκο πια αυτό το πακέτο, γιατί είναι λίγο προβληματική η ιστορία. Και η βασική επίκριση είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα κλαδικά, τομεακά, γιατί πρόκειται για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων με διαφορετικά δικαιώματα και διαφορετική έτσι, μεταχείριση. Μπορεί να είναι στόχος της οδηγίας η απλούστευση, η απλοποίηση των κανόνων δηλαδή και η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Αλλά κινδυνεύει να χαθεί αυτός ο στόχος με αυτή την κλαδική προσέγγιση. Τουλάχιστον εγώ δεν καταλαβαίνω τι απλοποιείται όταν έρχονται εργαζόμενοι στην ίδια επιχείρηση από διάφορες οδούς και διάφορους διάβλους. Έχουμε μπλε κάρτες, έχουμε άλλους εργαζομένους χωρίς τέτοια κάρτα, έχουμε αποσπασμένους, μετακινούμενους, ενδοεπιχειρησιακούς, ε, άλλους. Έχουμε εργαζομένους στην ίδια επιχείρηση με διαφορετικά καθεστώτα. Επιστήμονες, ερευνητές και κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή την απλοποίηση που είναι ο στόχος μας. Και ε, περιπλέκονται τα πράγματα αντί να απλοποιούνται. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων που έχουν ακριβώς αυτή την ειδίκευση και την εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο. Αυτό μας ενδιαφέρει να έχουμε ειδικευμένους εργαζόμενους και όσο περισσότερο κυκλοφορεί η ε, ε, εργατική, το εργατικό δυναμικό, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έχουμε. Ο κύριος Γιακολίνο λέει ότι χρειάζονται ακόμα κάποιες διευκρινήσεις στην οδηγία, παραμένουν ζητήματα σε εκκρεμότητα και για μένα ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι το εξής. Θα δημιουργηθεί μια αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ή δύο στα δύο ή δεν ξέρω, δύο χρόνων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στην αγορά εργασίας. Δεν θα ήταν σωστό. Επίσης νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση δεν με οδηγεί ε, αμυγός ε, μετανάστευσης ε, ή μετακίνησης. Είναι και ένα θέμα απασχόλησης. Έχει αντίκτυπο και στην απασχόληση. Τώρα δεν ξέρω μεγάλο ή μικρό, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, καλό θα ήταν η νομική βάση να ξεκαθαριστεί και να είναι και το άρθρο 153α που ασχολείται με την ασφάλεια και την υγιεινή συνεργασία με τους ε, όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και τέτοια θέματα εργατικά και εργασιακά και για εκείνους που έρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες. Έγινε λόγος και για τους ορισμούς προηγουμένως. Είναι σχετικά μεγάλη η συμφωνία εδώ και σχεδόν ομόφωνα όλοι θεωρούμε ότι θα πρέπει ορισμοί να είναι ακριβείς. Πώς ορίζονται τα στελέχη μιας επιχείρησης, τα διευθυντικά στελέχη, εμπειρογνώμονες κτλ. Και τι θα πει αν κάνουν knowledge, τι έχουν ειδικέ γνώσεις, εξαιρετικές γνώσεις. Πώς ορίζεται αυτό, χωράει και πολύ μεγάλη ερμηνεία. Παράδειγμα, σε μία κρόαση είπε κάποιος στη Γερμανία του Οργανισμού Απασχόλησης ότι ένας ειδικευμένο ε, ελεοχρωματιστής μπορεί να θεωρήσει ότι είναι εμπειρογνώμων και ειδικό ε, γιατί είναι τόσο χαλαρός ο ορισμός. Ε, ε διερωτώ με λοιπόν, αφού μιλούμε για απλοποίηση, χρειαζόμαστε ένα σωρό ορισμούς για το τι είστε ειδικό ή εμπειρογνώμων. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ήδη, ας πούμε στη βιβλία κάρτα, ε, ορισμό. Χρειάζεται τώρα καινούριο ορισμό η οδηγία αυτή. Μπορεί στη βλεκαρτα είναι διαφορετική η οδηγια το πεδίο εφαρμογής, αλλά η ομάδα εργαζομένων στην οποία αναφέρονται είναι η ίδια. Ε, οι εργαζόμενοι με μεγάλη δίκευση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ε, τους ορισμούς της πλεκάρτας. Κάτι άλλο που ακούσαμε στις ακροάσεις είναι το εξής. Κυκλοφορεί μια υποψία ως προς την έννοια των ε, ενδοεπιχειρησιακών ε, μετακινούμενων εργαζομένων. Το λέω αυτό γιατί έχω διατελέσει υπουργό εργασία στη Φιλανδία. Έχω εργαστεί και για την εκπόνηση αυτού του κειμένου. Αλλά αργότερα διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ακόμα δυναμίε και ελλείψεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότησε γι' αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι δεν είναι μου να χρησιμοποιούμε ε, αυτό τον ορισμό των μετακινούμενων ε, εργαζομένων ή των αποσπασμένων. Επίσης λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο ευνοϊκούς ε, κανόνες και ρυθμίσεις για τους ενδοεπιχειρησιακούς εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση με τους απεσπασμένους. Διερωτώ με το δικαστήριο πώς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. διότι η οδηγία αυτή δεν είναι στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, είναι στο μέγιστο. Επίσης, μέσω της οδηγίας αυτής ε, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες θα ε, έχουν τη δυνατότητα να έρχονται και να εργάζονται στην Ένωση για μία τριετία θα ήταν καλύτερο να ισχύει και για εκείνους η ίδια νομοθεσία με την νομοθεσία που ισχύει ε, για τους ντόπιου εργαζόμενους. Υπήρξαν πολλές δυσκολίες ε, στην εφαρμογή της οδηγίας για τους ε, απεσπασμένους εργαζόμενους και δεν νομίζω ότι θα μας διευκόλυνε να το κάνουμε και σε αυτή την οδηγία έτσι. Μάλλον θα και τα πράγματα. Γι' αυτό η δική μου Επιτροπή Απασχόλησης τονίζει την αρχή ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υφίστανται παντού την ίδια μεταχείριση, να ισχύουν παντού οι ίδιοι κανόνες ανεξαρτήτως προελεύσεως. Οι ίδιες συνθήκες εργασίας, συστήματα των κρατών μελών να ισχύουν. Και πάλι θα ήθελα να τονίσω ότι η οδηγία αυτή είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική και επαναλαμβάνω ότι είχαμε μια πάρα πολύ γόνιμη συνεργασία με τον κύριο Ιακολίνο και τους κοιόδης ηγητές της Επιτροπής Ελευθεριών αλλά και της Επιτροπής Απασχόλησης και θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω να ασχοληθούμε με τα αδύναμα σημεία ε, της οδηγίας για να τα ενισχύσουμε και να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Και θα πρέπει να ξέρουμε σε τι αποσκοπούμε. Οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να μετακινούν τους εργαζομένους τους, ωραία, να έχουν εργαζομένους που να έρχονται εδώ, χωρίς όμως αυτό να παραβιάζει ε, το καθεστώς και τα δικαιώματα των ντόπιων εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Now Βλέπω ότι μόνο ένας έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μπρόνς ή μάλλον και ο κύριος Μιλντερ. Άρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Πρώτα ο κύριος Μιλντερ, Έρνστ και τέλος ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Η φιλελεύθεροι είναι υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τις επιδοκιμάζουμε ως ένα επιπλέον βήμα προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και της κοινή μας πολιτικής για τη μετανάστευση και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης. Και είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Γιακολίνα για τις προσπάθειές του για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ήταν και καλή ακρόση και πολλαπλέ επαφέ που είχαμε για συνεννόηση. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Γιακολίνου. Βέβαια και οι φιλελεύθεροι έχουμε κάποιε ανησυχίε για του ασκούμενου. Γιατί αν έχουμε σε ένα κρατό ανεργία 25% και ένα πτυχιούχο ε, φεύγει. Καλό θα είναι να μπορούμε ε, όταν εμείς δεν μπορούμε να ε, καλύψουμε τις ανάγκες των πτυχίουχων μας και δεν μπορούμε να τους απασχολήσουμε, δεν ξέρω πόσο σκόπιμο είναι να δεχόμαστε αποφύτους ε, άλλων χωρών. Είναι καλή από αυτήν την άποψη η πρόταση για κολλήνωση ό,τι αφορά τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να διχάνουν ίσως με τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Και αν εκδίδεται άδεια παραμονής για κάποιον που θα έρθει να εργαστεί στην Ευρώπη, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα μέλη της οικογένειάς του. Δηλαδή να ανοίγουμε τις αγκάλες μας και προς αυτούς και να διευκολύνουμε την έκδοση αδειών παραμονής και για τα μέλη της οικογένειας. Τώρα, πριν την είσοδο στην Ευρώπη, ποια διάρκεια θα πρέπει να προκρίνεται ως ε, διάρκεια εργασία 12 μήνες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξάμεινο ο κύριος Γιακολίνο, θα περιμέναμε τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να στηρίζουν αυτό το δωδεκάμινο. Γιατί όποια, και όποια περίοδο και αν επιλέξουμε είναι πάντα συζητήσιμο ποια είναι η ιδανική, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στο δωδεκάμινο. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των διαφόρων κατηγοριών, νομίζω ότι η εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης μας το εξήγησε συζητήσιμα είναι ούτω ή άλλω όλα αυτά γιατί κατηγορηματικοί ορισμοί είναι δύσκολο να βρεθούν. Πάντως δεν είμαι κατά των προτάσεων για κολλήνο. Αλλά έχω αμφιβολίε για το κατά πόσο είναι σκόπιμο να επισέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ο κύριο Γιακολίνο προτείνει και κάποιε κάποιες για το μισθό αποσπασμένο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα πολιτικής της συγκεκριμένης επιχείρησης και είναι δύσκολο για οποιαδήποτε, επιχείρηση, ε, ε, ε, οποιαδήποτε κυβέρνηση ή κράτος μέλος να πει ότι αν κάποιος, κάποια επιχείρηση στέλνει υπάλληλό της στην Ευρώπη θα πρέπει ο μισθός του να είναι συγκεκριμένος. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του εργαζόμενου και της επιχείρησής του. Δεν μπορεί να επιβληθεί από τα κράτη της κυβερνήσης. Τώρα σε ό,τι αφορά την ομοιότητα αυτού του μισθού με τον ευρωπαϊκό μισθό εξαρτάται από το πεδίο δραστηριοτήτων ίσω επιχείρηση. Αλλά δεν νομίζω ότι ε, είναι αρμοδιότητα τη κυβέρνηση να προσδιορίσει το ύψο αυτού του μισθού που θα λαμβάνει αποσπασμένο. Η κυρία ε, Ευχαριστώ πολύ ε, τον εισηγητή. Νομίζω ότι στον κύκλο των σκιωδών ε, εισηγητών θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα σε βάθος γιατί χρειάζεται. Πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι θεωρώ σημαντικό καταρχάς να καθίσουμε να σκεφτούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη έχουμε ένα κατακαιρματισμό. Ε, τρόπο έχουμε κατηγορίες ή τάξεις εργαζομένων με διαφορετικά δικαιώματα, ε, με διαφορετικά νομικά πλαίσια και ε, προϋποθέσεις για την απασχόλησή τους για την εργασία που καλούν να κάνουν και με όλα τα συμπαραμαρτούντα. Ένα τεράστιο δίκτυο λοιπόν πολύ διαφορετικών ε, νομικών καθεστώτων και είναι και μεγάλο πρόβλημα προφανώς αυτό. Όχι μόνο για το πώς ε, το χειρίζονται τα κράτη-μέλη και οι εταιρείε, αλλά πώς το χειρίζονται και οι εργαζόμενοι. Πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε από νομικό πλαίσιο εννοώ, από νομικούς κανόνες και τι δεν χρειαζόμαστε, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ζητάμε και τι θέλουμε και τι κανόνες έχουμε. Θέλω να γίνει αυτή η συζήτηση, παρακαλώ, σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών μαζί με τον εισηγητή μας. Ένα δεύτερο. Είναι βέβαια πάντα το θέμα των ορισμών. Η ακρόαση έδειξε πόσο εκρηκτική είναι αυτή η οδηγία, το σχέδιο οδηγίας και οι εκθέσεις που συνδέονται μαζί της. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος είναι αυτός ο ειδικό εργαζόμενος που θα έχει τις σούπερ γνώσεις και τα φοβερά προσόντα και τα λοιπά, ο καταπληκτικός, δεν έχω καταλάβει. Ε, ούτε από την έκθεση είναι σαφές αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι, ποιοι είναι οι σούπερ ε, σπεσιαλίστες με τις τρομερές γνώσεις που φέρνουμε. Ε, μπορούμε να το οροπήσουμε όπως θέλετε με καλολογικά στοιχεία, αλλά δεν ευσταθεί νομικά. Ούτε είναι σαφές τι εννοούμε. Και στην ακρόαση επίσης φάνηκε ότι ο όρος όμιλος, concern, είναι επίσης τελείως θολός και ασαφής. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Και το τελευταίο, η συμμεταχείριση με τους ε, ε, χώριους εργαζομένους, να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά και αυτό πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη δηλαδή. Ποια θα είναι τα δικαιώματά τους, τα κοινωνικά, ε, τα εργασιακά, με τις οικογένειες τους τι γίνεται, θα τους παίρνουν οι πολυεθνικές και θα τους πηγαίνουν από εδώ εκεί, τι θα τους κάνουν. Όλα αυτά χρειάζονται πολύ μεγάλη καθάριση και έχω πάρα πολύ ανάμεικτα συναισθήματα για την έκθεση γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Οι ενδοεπιχειρησιακές αποσπάσεις μας αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της οικονομικής μετανάστευσης δεν μιλούμε για τις ανθρώπινες φιλοδοξίες, ε, ε τις επαγγελματικέ, αλλά ε, ικανοποιούμε περισσότερο τις ε, ανάγκες των μεγάλων πολυεθνικών. Ακούσαμε το πρωί για την ανάγκη των, της αγοράς εργασίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μία αγορά είναι ε, ένας τρόπο όπου έχουμε αγοραπολισίες αγαθών, εμπορευμάτων, όχι ανθρώπων. Εδώ μιλούμε για ανθρώπινους πόρους, αν ήταν ανώνυμα τμήματα της παραγωγής, ανώνυμα γρανάζια της παραγωγής οι άνθρωποι και όχι έμψυχα όντα. Υποτίθεται ότι θέλουμε να ε, ε, ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πολιτών, των ανθρώπων, όχι τις ανάγκες των ε, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενώ αυτό κάνουμε φαίνεται εδώ. Εδώ βέβαια μιλούμε για αποσπάσεις ε, στελεχών, επαγγελματιών, εμπειρογνωμών από τρίτες χώρες. Και όταν λέμε τρίτε χώρε, εννοούμε πολύ συχνά χώρε του τρίτου κόσμου. Πολλοί από αυτού του ανθρώπου ε, εκπαιδεύτηκαν και καταρτίστηκαν με ελάχιστου πόρου. Και ε, γίνεται ένα κυνήγι κεφαλών, όπω λέμε, ε, προκειμένου να απασχοληθούν στον αναπτυσσόμενο, στον αναπτυγμένο μάλλον κόσμο. ακούσαμε ένα εκπρόσωπο του Μάλι πριν από λίγε μέρε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πέσει την προσοχή μα το υψηλό ποσοστό στις ε, δεκαετία του 30 ε, πτυχίουχων του Μαλή που εργάζονται στην Αλοδαπή, κυρίω σε ανεπτυγμένε χώρε. Νομίζω ότι για την ανάπτυξη αυτών των χωρών, και ελπίζω να μην ακούγεται απεσιόδοξο, ε, το καλύτερο είναι να επενδύσει στους πιο ταλαντούχους πολίτες. Αν μεταφέρονται αυτοί οι ταλαντούχοι προς τι ανεπτυγμένε αναπτυγμένες χώρες, τότε είναι που θα καταδικάσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες σε αιώνια ένδια και στασιμότητα. Αν θέλουμε να τις βοηθήσουμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τα εκπαιδευτικά του συστήματα για καλύτερη εκπαίδευση. Επίσης, τα κράτη θα πρέπει να κρατήσουν τον έλεγχο των συνόρων τους και να μην ε, εκχωρούν τις αρμοδιότητές τους σε αρπακτικές και άπλιστες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ, η ε, Σας ευχαριστώ. Ακούγοντας τον προ... τους προλαλήσαντες και κυρίως τον εισηγητή μας φυσικά, αρχίζω και προβληματίζομαι. Τι ακριβώς επιδιώκουμε με την οδηγία αυτή. Θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα από τα κέρια ζητήματα. Το θέμα το μισθολογικό, το μισθό ενός αποσπασμένου ενδοεπιχειρησιακά που εργάζεται στην Ευρώπη. Ο εισηγητής προτείνει σε μια τροπολογία ότι ο αποσπασμένος αυτός θα πρέπει να κερδίζει τον ίδιο ή παρόμοιο μισθό με έναν ε, Ευρωπαίο εργαζόμενο σε αντίστοιχο επάγγελμα. Όταν όμως κανείς ε, προέρχεται από μια χώρα με πολύ χαμηλότερους μισθούς είναι λογικό και ε, κατανοητό να ζητούμε κάτι τέτοιο. Γιατί φοβόμαστε μήπως οι αποσπασμένοι περιθωριοποιήσουν τους ε, Ευρωπαίους εργαζόμενους ή αποσπασμένους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τους εκτοπίσουν από την αγορά εργασίας. Όμως κάποιος προέρχεται από την Αραβική Χερσόνησο ή από τον Καναδά ως αποσπασμένος στην Ευρώπη, τότε θα ήταν πολύ περίεργο αυτό το αίτημα για ισότητα με, ε, τον ευρωπαϊκό αντίστοιχο μισθό. Θα πρέπει όμως να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει και δεν μπορούμε να το επιλύσουμε καν με την οδηγία αυτή, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να το εντοπίσουμε και να το αναγνωρίσουμε. Είναι ακριβώς επειδή η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους δεν ε, ε διαθέτησε ικανοποιητικά το θέμα των μισθών, δεν μπορούμε από αυτή την άποψη να κάνουμε χειρότερη την οδηγία για τις αποσπάσεις ενδοεπιχειρησιακά. Δεν είναι ισότητα μεταχείριση αν οι αποσπασμένοι αυτοί ε, ενδοεπιχειρησιακά ε, τύχουν οι μεταχειρήσει με του αποσπασμένου. Επειδή ακριβώ οι αποσπασμένοι ε, έχουν ελάχιστα δικαιώματα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε εξομοίωση προ τα κάτω. Χαίρομαι για τη διευκρίνηση των δικαιωμάτων των μελών των οικογενειών αυτών των αποσπασμένων εντός μιας επιχείρησης. Είναι σημαντικό να επιτρέπουμε ε, στους εργαζόμενους αυτούς να εργαστούν στη χώρα υποδοχής και γίνεται πιο ελκυστική αυτή η προσφορά εφόσον επιτρέπουμε και στις οικογένειές τους να μεταναστεύσουν. Βέβαια, σε αυτούς τις εποχές ε, της χειραφέτησης ε, θα ήταν κάπως ε, περίεργο να αφήνουμε να περιορίζουμε τα μέλη της οικογένειας, να τους περιορίζουμε κατοίκον ουσιαστικά, να κάθονται στο σπίτι δηλαδή και να μην κάνουν τίποτα. Ο κύριος Ιακολίνο μίλησε και για θέματα μετανάστευσης και ένταξης κοινωνικής. Όταν μιλούμε όμως για αποσπάσεις εντός μιας επιχειρήσης, δεν νομίζω ότι η ένταξη είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, η κοινωνική ένταξη. Γιατί ο αποσπασμένος αυτός συνήθως έχει και σύμβαση που προβλέπει και παλινόστηση, παλινόστηση του. Πολλά αναφέρθηκαν για το θέμα αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να οργανώσουμε ξεχωριστή συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών για να τα εξετάσουμε όλα αυτά και μάλιστα σχετικά σύντομα. Ο κύριος Μωράς ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπριγκεβιτσούτε, η σκιώδη συγγήτρια των Σοσιαλιστών, συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόληση. γι' αυτό αποσιάζει. Ήθελε να εξετάσει το ζήτημα της ε, ίσης μεταχείρισης. Μας το ανέφερε η κυρία Γεκοσάρη, το θέμα του ορισμού των ε, ψηλών στελεχών με εξαιρετικέ γνώσεις, το θέμα των ασκουμένων, το θέμα της ε, οικογενειακής επανένωσης και ποια θα είναι ακριβώς η εμβέλεια αυτού του θέματος στην οδηγία αυτή για τις αποσπάσεις εντός μιας επιχείρησης. Δεν θέλω να προεξοφλήσω τη θέση ε, της Κιόδους απλώς ε, θα ήθελα να επισημάνω εκ μέρου αυτά τα σημαντικά θέματα, που σίγουρα φαντάζομαι θα θυγούν, και στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Επανέρχομαι τώρα στον κύριο Τζακολίνο, τον εισηγητή μας, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Άκουσα όλες τις ε, παρεμβάσεις ε, με μεγάλο ενδιαφέρον και θα σχολιάσω εντάχει, αρχίζοντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναφέρθηκε στην ε, συνεργασία από όπου προέκυψαν ορισμένες διορθώσεις, διορθώσεις των ορισμών. Επί του θέματος ε, εργαζόμαστε τώρα, επ' αυτού του θέματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Προεδρία για αυτή την πολύ καλή συνεργασία γιατί θα πρέπει να φτάσουμε σε έναν εξισορροπημένο σε έναν ισορροπημένο ορισμό του άρθρου 16 και σε σχέση με την κινητικότητα σε όσον αφορά τις ενδοεπιχειρησιακές αποσπάσεις η περίοδος αναφοράς μειώνεται από 12 σε 6 μήνες. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να επέλθουν και άλλες μικροαλλαγές για την ολοκλήρωση του πλαισίου. Υπάρχει και μία τροπολογία επ' αυτού και νομίζω ότι η συνεργασία βαίνει καλώς. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Γιακονσάρη, η οποία μίλησε για την αγαστή συνεργασία που ε, υπάρχει με τους σκιώδεις. Ήδη έγινε μία συνάντηση λίγες ε, μέρες πριν και προβλέπονται και άλλες συναντήσεις. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις παρόλα αυτά. Πρόκειται για μία οδηγία για την νόμιμη μετανάστευση, αλλά σχετίζεται με την αγορά εργασίας όπου μιλάμε για ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι συμβατικές σχέσεις και ιδιαίτερα πόσο καιρό πρέπει να, να έχει απασχοληθεί ο εργαζόμενος πριν να μπορέσει να αποσπαστεί σε μια τρίτη χώρα. Εμείς προβλέπουμε μια τροπολογία που αναφερόταν στους 12 μήνες, τώρα μιλάμε για 6 μήνες. Θα πρέπει να πρόκειται για έναν εργαζόμενο που τουλάχιστον για 6 μήνες αδιαλείπτος έχει εργαστεί στην επιχείρηση. Αυτό μου φαίνεται απόλυτα λογικό. Επίσης, όπως είπε και η κυρία Γιακονσάρη, θα πρέπει να αναφερθούμε στις διευκολύνσεις για την οικογένεια μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης ισορροπίας. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ενιαία άδεια παραμονής και εργασίας ή κατά πόσο θα πρέπει να προβλέψουμε την επανένωση της ε, οικογένειας ως προς τις αμοιβές η συνάδελφος ε, Σαρζεντίνη αναφέρθηκε επί του θέματος, καθώς και ο συνάδελφος ε, Μωράης. Στην προγενέστερή μου δραστηριότητα ήμουν διευθυντής ε, μίας επιχείρησης με 6.000 εργαζόμενους. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι μπορούν να έχουν διαφορετικό συμβατικό ε, πλαίσιο και διαφορετικές συμβάσεις τη στιγμή που επιτελούν την ίδια εργασία, αυτό μου φαίνεται παράλογο. Το θέμα των ορισμών είναι πολύ σημαντικό, όπως προελέχθη. Αλλά αν δείτε τις ε, τροπολογίες που υπέβαλα, βλέπετε ότι οι οδηγίες αναφέρονται στο γεγονός ότι το διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να έχει ιεραρχικά προσόντα, θα πρέπει να έχει ε, συγκεκριμένες, να πληρεί συγκεκριμένες παραμέτρους οι οποίες να είναι μετρήσιμες ενώ απαντώντας στον κύριο Μίλτερ αναφερόμενος στους ασκούμενους υπάρχει κοινοτικό προτιμησιακό καθεστώς όπως φαίνεται και από την πρώτη μου τροπολογία έτσι ώστε να αλλάξει η αιτιολογική σκέψη 8 διότι η σταζιγέρ από τρίτες χώρες, ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τον ε, αριθμό αυτών που προέρχονται από τα κράτη-μέλη, των ασκουμένων που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Επίσης, ως προς την εξειδίκευση, μιλήσαμε για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και αυτό εξαρτάται από το πόσο, πώς θα ορίσουμε τις, οδηγίε, τις οδηγίες συγγνώμη, ε, και τους ορισμούς. Τι θέλουμε, ποιον θέλουμε το άρθρο 8, κυρώσεις. Θα πρέπει να προβλέψουμε συγκεκριμένες κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ε, θα πρέπει να έχουμε μία απλουστευμένη συνεργασία και εφαρμογή, όπως είπε η κυρία Γιακονσάρη οικογένεια. Βασική έννοια η οποία ε, προβλέπεται μέσα στα πλαίσια της επανένωσης της οικογένειας. Και μετά υπάρχει και το θέμα της κινητικότητας, το άρθρο, το περίφημο άρθρο 16. Τι θα γίνει με έναν εργαζόμενο που προέρχεται από την Ινδία και αποσπάται στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ιταλία. Το θέμα αυτό παρουσιάζει προβλήματα και οι συνάδελφοι που παρενέβησαν μπορούν να συνεισφέρουν διότι ο κύριος Μπρόνς είπε ότι μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά, να αξιοποιήσουμε διότι το 21% των νέων δεν εργάζονται. Στην Ιταλία πρόκειται για το 28%. Το θέμα είναι κοινό λοιπόν και είμαι πεπισμένος ότι κατά την προσεχή συνάντηση με τους σκιώδεις ο, κανένας, ο καθένας θα μπορέσει να συνεισφέρει. Και προτείνω πρόεδρε να ορίσουμε ως προθεσμία υποβολής τροπολογιών την 12η Ιουλίου έτσι ώστε ο καθένας και η κάθε πολιτική ομάδα να μπορέσει να εκφράσει τις απόψεις της. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, Πρόεδρε. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Κυρία Γιακουνσάρη, πολύ σύντομα από την Επιτροπή Απασχόλησης, διότι έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μιλήσαμε για την διαφυγή, ε, διαρροή εγκεφάλων. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει, δηλαδή θα πρέπει να, έχουμε, να αποφύγουμε αυτή τη διαρροή. Πρόκειται για μία περίοδο εργασίας που επεκτείνεται σε τρία χρόνια ως προς την ίση μεταχείριση. Πού βρίσκονται οι, πιο, οι μηχανικοί που στοιχίζουν πιο φτηνά παγκοσμίω. Πολλοί πιστεύουν στην Κίνα. Ε, παλαιότερα πιστεύαμε στην Ουκρανία, ότι βρίσκονται στην Ουκρανία. Εγώ νομίζω ότι αν μια φιλανδική-γερμανική επιχείρηση θέλει να προσλάβει μηχανικούς από τρίτες χώρες για να αποφευχθεί το μισθολογικό dumping, τότε δεν θα τους προσλάβουν επειδή έχουν χαμηλότερο μισθό, αλλά επειδή θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους. Αυτό που τους ενδιαφέρει λοιπόν είναι να προσλάβουν Ισπανούς, Πορτογάλους ή Πολωνούς μηχανικούς. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, να μην έχουμε μια, ε, μια διπλή αγορά εργασίας. Γι' αυτό η συμμεταχείριση έχει μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ όλους. Ωραία, εδώ σταματάμε και λαμβάνουμε υπόψη τις υποδείξεις, υποβολή τροπολογιών, λοιπόν προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 12 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. 12 Ιουλίου ημέρα Τρίτη μέχρι τις 12 το μεσημέρι για τροπολογίες επί της έκθεσης για κολίνο. Ως προς την Επιτροπή Αποασχόλησης, νομίζω ότι η προθεσμία που ορίστηκε είναι για τις 22 Ιουνίου. Έτσι δεν είναι η κυρία Γιακονσάρη για τα άρθρα που αποτελούν δικαιοδοσία της Επιτροπής Απασχόλησης δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού. Ωραία, προχωράμε τώρα με καθυστέρηση και προχωράμε στο σημείο 21 που αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών μέσα στα πλαίσια της εποχικής απασχόλησης ο κύριος Σέρτζο Κοφεράτη είναι από κοινού εισηγητής και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να λάβουμε υπόψη το σχέδιο έκθεσης ε, του εισηγητή της Επιτροπής Λίμπε, του κυρίου Μωράης και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοφεράτη για να μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης. Ο κύριος Μωράης είναι υπεύθυνο για το θέμα των εποχικών απασχολουμένων και μετά την ακρόαση που διοργανώθηκε τον Απρίλιο θα πρέπει να ορίσουμε μία ημερομηνία για υποβολή τροπολογιών. Ας ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Μωράης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι στη συζήτηση την προηγούμενη οδηγία ε, των ενδοεπιχειρησιακών αποσπάσεων είδαμε πόσο περίπλοκος είναι ο κλάδος ε, αυτός. Είναι τρεις φάκελοι που αφορούν μετανάστευση, μετακίνηση εργαζομένων, ε, τομεακά, τρία διαφορετικά θέματα τι ε, προσπαθούμε. Και με τη γαλάζια, την μπλε κάρτα πριν τη Λισαβόνα, έχουμε θεσπίσει ένα καθεστώς ημιμόνιμης απασχόλησης. Είναι ε, αυτή η υπόθεση που μας απασχολεί τώρα, η ε, αποχειακή απασχόληση. Πολλές ανησυχίες συνδέονται με αυτό και εκφράστηκαν και κυρίως το θέμα της που βέβαια είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης. Τώρα που βρισκόμαστε χρειάζεται βελτίωση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά οι προτάσεις για αυτό το θέμα. Και τι προσπάθησα εγώ να κάνω. Να βεβαιωθώ ότι ασχολούμαστε και με θέματα εκμετάλλευσης που είναι υπαρκτά και να ε, μειώσουμε την ανάγκη για ε, έκτακτη απασχόληση, ε, για αντικανονική ανώμαλη απασχόληση. Είναι η εποχιακή απασχόληση ένα γεγονός, εποχιακό μεν αλλά μόνιμο που επανέρχεται. Δεν υπάρχει λόγος να θεωρείται κάτι έκτακτο. Και κάτι ε, που δεν συζητούμε δημόσια είναι το πεδίο εφαρμογής που είναι αρκετά περιορισμένο. Διαφέρει από το προηγούμενο θέμα της ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης γιατί συμπεριλαμβάνει και ανειδίκευτούς εργαζομένους εδώ αλλά είναι συγκεκριμένη κατηγορία που ήδη έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά και ξανά. Η προσέγγιση είναι κομμένη και ραμμένη ε, στα μέτρα των όσων ακούσαμε στην ακρόαση τον Απρίλιο, αλλά είχαμε και εκτενέστατες συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, με πάσης φύσεως ε, φορείς, όχι μόνο επειδή συζητούσαμε την ενιαία άδεια, αλλά προσπαθούσαμε να διδαχθούμε και από την εμπειρία που έχουν εκείνοι και από τις προηγούμενες. Αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω με την πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν να διατηρήσω αυτά τα στοιχεία που θεωρώ κρίσιμα και σημαντικά. Από την αρχή της συζήτησης για την εποχιακή απασχόληση θα θυμούνται οι ε, συνάδελφοι ότι είχαν έρθει και τα Εθνικά Κοινοβούλια και μας είπαν ότι εδώ η επικουρικότητα είναι κομβική και τα λοιπά. Βεβαίω τα κράτη-μέλη, προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να είναι ε, απολύτως ε, κύρια των ε, αριθμών των εργαζομένων που επιθυμούν και προηγουμένως να έχουν ελέξει κατά πόσον οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από υπηκόους των χωρών τους ή πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν καταφύγουν στους εποχιακούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να μειωθεί η άτυπη εργασία και να αυξηθούν όμως και τα κίνητρα επιστροφής των εποχικών εργαζομένων που έρχονται στην Ένωση στις χώρες τους. Έρχονται σε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας και μετά φεύγουν. Και το θέμα δεν είναι να αφαιρέσουμε αυτούς τους εργαζομένους από τις χώρες τους που τους χρειάζονται, γιατί έτσι πάει και χαμένη η αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε ε, ως κράτη-μέλη ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό λοιπόν εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους αυτούς ε, και είναι σημαντικό ε, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταλάβει ότι είναι κυκλική αυτή η μετανάσταση. Ιδιαίτερα το άρθρο 12 ορίζει ότι όσοι δεν ε, συμμορφώνονται προς την υποχρέωση επαναπρατισμού τους όταν λύγει η άδειά τους να μην έχουν τη δυνατότητα να επανέρχονται την επόμενη ε, χρονιά. Επίσης το άρθρο 12 ε, λέει ότι μπορούν να ζητήσουν και πολυετή άδεια, δηλαδή να μπορούν να έρχονται την επόμενη χρονιά, που αυτό είναι επιπλέον κίνητρο ακριβώς για να τηρούν την υποχρέωση επιστροφής στις χώρες τους. Βεβαίως, το θέμα της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβή είναι αποκλειστικότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη της Επιτροπής Απασχόλησης, ε, το συντάξει εκεί για την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε. Μετά τη Σοχόλμη και τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, είναι ένα θέμα που αφορά και την Επιτροπή μας, αλλά και την Επιτροπή Απασχόλησης. Γι' αυτό υπάρχουν ορισμένες ε, ε, αποκλειστικές αρμοδιότητες και ορισμένες συντρέχουσες δική μας με τις Επιτροπές Απασχόλησης. Το θέμα λοιπόν της αμοιβή είναι θέμα της Επιτροπής Απασχόλησης αποκλειστικά, αλλά καλό είναι που το συζητάμε και εμείς εδώ στην Επιτροπή Ελευθεριών, γιατί σε πρακτικό επίπεδο βασικά δεν θέλουμε να έχουμε ε, ομάδες εργαζομένων ε, που έρχονται να υπονομεύουν την κατάσταση την εργασιακή των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η, ίση, η μεταχείριση ίση είναι βασικό στοιχείο και νομίζω ότι και ε, οι δύο επιτροπές έχουν εκφραστεί στο παρελθόν. Το θέμα τώρα της διάρκειας της παραμονής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το πολύ έξι μήνες. Το διατηρώ εγώ στην έκθεσή μου και πάλι Μπορούμε να συζητήσουμε ε, ό,τι θέλετε. Εγώ προτίμησα να τήρησω το εξάμεινο της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε σχέση με τη στέγη τώρα. Πώς θα τους προστατεύουμε από την εκμετάλλευση, τους εποχιακούς εργαζομένους. Το ξέρουμε ότι ε, σε πολλές χώρες είναι πολύ καλό το επίπεδο αξιοπρεπές, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπου το επίπεδο δεν είναι ε, ούτε ίσο ούτε αξιοπρεπές. Το θέμα της στέγασης τους είναι πάρα πολύ περίπλοκο, γιατί από τη μια θέλουμε να έχουμε αξιοπρεπείς και σωστές ε, συνθήκες για εποχιακούς εργαζομένους που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σκλάβοι άνθρωποι, θα πρέπει να εργάζονται κανονικά και είναι θέμα και των κοινωνικών εταίρων αυτό και των κρατών μελών. Γιατί όταν ε, έχουμε μια ομάδα εργαζομένων που ζουν σε φρικτές συνθήκες και τη χάνουν τέτοιες μεταχείρισεις είναι κακό για όλη την κοινωνία. Ε, το θέμα με τους εποχικούς εργαζομένους είναι ότι θα πρέπει να ζουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και αυτό επίσης έχει κοινωνικές επιπτώσεις. Καλή ελαστικότητα, αλλά θα πρέπει να πούμε ποιο είναι το σε βιωτικό επίπεδο. Ε, ως ορισμός είναι δύσκολο αυτό να βρεθεί. Υπάρχει μια επιτροπή του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα που κάπως το ορίζει αυτό και έχουμε βάλει και στην έκθεση την ιδέα ότι οι εποχικοί αυτοί εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να τη χάνουν εκμετάλλευση βεβαίως ε, και όταν συζητάμε αυτά τα θέματα μπαίνουμε σε χωράφια ε, ελευθεριών και των εργοδοτών που θέλουν να έχουν ελαστικότητα και ελευθερία κινήσεων αλλά Το θέμα είναι να έρχονται αυτοί να, εργάζονται, να βοηθούν την αγορά εργασίας μας, αλλά με τα εμβάσματά τους και το συνάλλαγμα που στέλνουν να βοηθούν και την ε, οικογένειά τους και τη χώρα τους. Αλλά να έχουν και αξιοπρεπείς και σωστές συνθήκες διαβίωσης. Αυτό μας αφορά και εμάς. γιατί το έχουμε συζητήσει και σε επισκέψεις και αποστόλες που είχαμε κάνει. Τώρα, σε ποιο πεδίο θα εφαρμοστεί η οδηγία. Ε, κλαδικά το συζήτησα με τους κοινωνικούς εταίρους και με πολλούς και είπαμε ότι να ασχοληθούμε με τη γεωργία, την ανθοκομία και τον τουρισμό. Αυτοί είναι οι τρεις τομείς που απασχολούν κυρίως εποχικούς εργαζομένους. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που δεν συμπεριλαμβάνουν εδώ κλάδι της οικονομίας, αλλά ε, ο τρόπος ε, που επέλεξα να κάνω την έκθεσή μου για την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτός. Ότι θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις εκτός αυτών που σας ανέφερα που απασχολούν εποχικούς εργαζομένους αλλά να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη αν θα επεκταθούν ε, και σε άλλους τομείς εκτός αυτών των τριών ε, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι τρεις είναι η γεωργία, η και ο τουρισμός. Αλλά είναι πραγματικά εποχή και επασχόληση και όχι καλυμμένη ε, άλλη τομής. Μετά υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις ε, και όταν δεν τηρούνται από τους εργοδότες θα πρέπει να συνοδεύουν και από Και είναι θεμητή ανάγκη ε, να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση εκμετάλλευσης ε, και προώθησης από κάποιους εργοδότες της παράνομης σε μαύρης εργασίας. Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι επιθεωρήσεις, παρακολουθείτε η κατάσταση. Επανειλημμένα ακούμε από τους κοινωνικούς εταίρους ότι η οδηγία θα είναι όσο αποτελεσματική είναι η έλεγχη και το σύστημα ελέγχων τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι θα γίνονται σωστοί έλεγχοι επιθεωρήσεις και θα έχουν αποτελέσματα. Τα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν την ίδια στάση παντού, να κάνουν πολύ καλές επιθεωρήσεις και ελέγχους, αλλά όχι. Τώρα, τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελιών και παραπώνων, γιατί ακούμε και τέτοια θα πρέπει να αποφευθεί η θυματοποίηση και να βοηθούν οι καταγγελίες και τα παράπονα για να ανέβει το επίπεδο παντού. Και ένα τελευταίο για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά πολίτες τρίτων χωρών που ζουν εκτός της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης όμως αντέδρασαν πολύ σφοδρά ορισμένοι συνάδελφοι. Είπαν ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια γέφυρα, ένα σύστημα σύνδεσης ορισμένων πολιτών τρίτων χωρών που ε, διαμένουν παράνομα στην Ένωση και επασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους ήδη. Εγώ πρότεινα μία διετία ως μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να βρεθεί κάποια ρύθμιση ε, για αυτούς τους εργαζομένους. Γιατί το κάνω αυτό. Και καταλαβαίνω ότι υπερβαίνει ενδεχομένω την ε, πρόταση, αλλά ακούστηκε στην ακρόση και νομίζω ότι θα πρέπει με τι άλλο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Συμπέρασμα. Έχουμε ένα τετελεσμένο σε κάποιους κλάδους της οικονομίας και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ακριβώς για να σπάσει η εκμετάλλευση. Καταλαβαίνουμε ότι η εποχική απασχόληση είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ένα μόνιμο στοιχείο κάθε χρόνο η εποχική απασχόληση της αγοράς εργασίας και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να φροντίσουν και τις οικογένειές τους με τα εμβάσματα που στέλνουν, με το συνάλλαγμά τους. Να το ε, ελέγξουν λοιπόν τα κράτη-μέλη, παραμένει στα χέρια των κρατών μελών αυτό και ελπίζω να ανέβει και το επίπεδο και οι προδιαγραφές και να σταθεροποιηθεί αυτός ο κλάδος της οικονομίας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, ακόμα και αν είναι εποχικός. Ευχαριστώ πολύ τους κοιόδης ηγητές, ε, κάναμε συνεδριάσεις, συνεργαστήκαμε. Το θέμα αυτό είναι ευαίσθητο και λεπτό από πολλές πλευρές. Ευχαριστώ λοιπόν τους κοιόδης ηγητές και ε, την κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου που ήταν συντάκτη γνωμοδότης της Επιτροπής Γυναικών. Την έστειλε πολύ νωρίς την γνωμοδότησή της. Ευχαριστώ. Thank you, Now we... Ευχαριστούμε, Κλοντ. Τώρα θα ακούσουμε σύντομα τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμά μας εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικότατη. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον εισηγητή σα για την αγαστή συνεργασία, την έκθεσή του και να πω ότι ένα στοιχείο που ήταν σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπέβαλε την έκθεση είναι φυσικά η προσπάθεια πλούστευση ε, της ε, υποδοχή τέτοιων εποχικών εργαζομένων, ώστε να ε, βρίσκονται εδώ όταν τους χρειάζονται οι εργοδότες. Και είπαμε ότι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που θέλαμε να καλύψουμε είναι η προστασία των ευάλωτων, πιο ευάλωτων ομάδων και να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευσή τους. Στις τροπολογίες που κατατέθηκαν για την έκθεση, αυτό το στοιχείο της προστασίας των ευάλωτων εργαζομένων έχει ενισχυθεί. Είμαστε υπέρ της πρόσβασης στην πληροφορία, στην ενημέρωση, μηχανισμός ε, υποβολής αιτιάσεων, παραπώνων κτλ. Ορισμένα στοιχεία διαφέρουν από την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο θέμα για το πεδίο εφαρμογής και την δυνατότητα για την ε, εφαρμογή σε ό,τι αφορά την επικράτεια ενός κράτους. Αυτή είναι μια δυνατότητα που υπάρχει όταν υποβάλλει κανείς την πρόταση. Αυτοί όμως είναι προσωρινοί μετανάστες, έρχονται για εποχική απασχόληση, για λίγους μήνες μόνο. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε σκόπιμο να εφαρμόσουμε μόνο αιτήσει, να δεχτούμε μόνο αιτήσει ε, για μετανάστες που περιλαμβάνονται στην ε, χώρα, από τη χώρα προέλευσης για να αποφευχθούν καταχρήσεις. Είναι πολύ προσωρινός ε, ο χαρακτήρας της διάρκειας, οπότε λόγω της προσωρινότητας αυτής δεν υπάρχει καν ανάγκη οικογενειακής επανένωσης. Yeah. Γιατί ίσως κάτι τέτοιο δημιουργούσε ευκαιρίες για κατάχρηση. Επίσης, ε, δεν καλύψαμε τη δυνατότητα, δεν καλύψαμε την πιθανότητα ε, των λάθρων μεταναστών. Η οδηγία αυτή αφορά τους ε, νόμιμα εργαζόμενους, τους νόμους μετανάστες. Και το θέμα της ε, επισημοποίησης είναι θέμα κράτους μέλους. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των εποχικών εργαζομένων, θέλησαμε ένα στελτικό ορισμό για είναι όντως εποχιακή απασχόληση. Βέβαια και ως προς την εποχιακότητα αυτή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε επαφείται στη διακριτική ευχαίρεια των μερών να αποφασίσουν ποιοι είναι οι τομείς για τους οποίους θα ισχύσει αυτή η πρόταση. Ένα άλλο θέμα είναι οι θεωρήσεις και οι άδειες. για τους εποχικά αποσχολούμενους που έρχονται για λιγότερο από τρίμηνο θα πρέπει να, έχουν, να είναι εφοδιασμένοι με θεώρηση Σέγγεν. Αυτούς που υπερβαίνουν το τετράμινο προτείνουμε άδεια. Βέβαια, τα κράτη-μέλη μπορούν από την αρχή να ζητήσουν άδεια και για συντομότερες διάρκειες. Πάντως το σημαντικό είναι να έχουν οι εποχικά απασχολούμενοι τα, όλοι ίδια δικαιώματα, ίσα δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το έγγραφο, αν θα είναι θεώρηση δηλαδή η διαμονή, αλλά να εξασφαλίζονται ίσα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και το εξάμεινο στο ημερολογιακό έτος, προτείναμε αυτή την περίοδο αναφοράς για να αποφύγουμε την επιβάρηση της ε, δημόσιας διοίκησης. Γιατί το μερολογιακό έτος ούτως ή άλλως είναι σημείο αναφοράς και για φορολογικά ζητήματα, γι' αυτό το θεωρήσαμε και δόκιμη αναφορά και για την περίπτωση αυτή τώρα να μεταβούμε από το ημερολογιακό έτος στο δωδεκάμινο. Νομίζω ότι αντιβαίνει, αντιστρετεύεται το στόχο της πρότασης που μιλάει για ένα εξάμηνο μέσα σε ένα δωδεκάμινο. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον όχι. Αν προτιμάτε το 12 μήνο δεν νομίζω ότι θα προσβληθεί ο σκοπό τη οδηγία. Οπότε αν το προτιμάτε από το ημερολογιακό έτο, δεν θα έχουμε αντίρρηση. Ό,τι αφορά την προστασία των ε, εποχιακά εργαζομένων επίση ε, είναι ένα σημαντικό θέμα. Τη δυνατότητα των εργοδοτών να καλύψουν ε, το κόστος μετάβαση ταξιδιού. Προσοχή όμως για να μην αποθαρρύνουμε έτσι με τέτοια έξοδα τους εργοδότες ε, από την ε, πρόσληψη, νόμιμη πρόσληψη μεταναστών από τρίτες χώρες για να μην επηρεάσει αρνητικά, να μην τους αποτρέψει αυτό το κόστος του ταξιδιού από την πρόσληψη. Αυτά και είμαστε στη διάθεσή σας ε, για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την περαιτέρω παροχή διευκρινήσεων. Η κυρία Βαλάση από την Ουγγρική Προεδρία, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι εξαιρετικά λακωνική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μωράες για την εξαιρετικά λεπτομεριακή έκθεση του και να πω εντάχει πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στα θέματα που δεν αναφέρθηκαν στην ακρόαση. Και η Ουγγρική Προεδρία θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο, αυτή την πρόταση και στη συζήτηση, στις διαβουλεύσεις ακούσαμε και εμπειρογνώμονες για κοινωνικά ζητήματα και πιστεύουμε ότι καταφέραμε τελικά να διευκρινίσουμε πολύ σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν και τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης, μιλήσαμε για εποχιακή απασχόληση που υπερβαίνει το τρίμηνο μέσα σε μια συνολική περίοδο εξαμήνου. Αυτό είναι αφισβητήσιμο ακόμη, είναι επίμαχο το θέμα, γιατί πολλές χώρες εξέφρασαν ανησυχία. ό,τι φορά το σχέδιο οδηγία και το θέμα της, του κώδικα θεωρήσεων και το κατά πόσο είναι συμβατά τα δύο μεταξύ τους. Αν μιλούμε για περίοδο που δεν υπερβαίνει το τρίμηνο, εδώ προβλέπεται υποχρεωτική αίτηση με βάση τους υφιστάμενους κανόνες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα και η συμμεταχείριση και για τους ε, εποχιακά απασχολούμενους. Αυτό όμως είναι σχετικά δευτερεύον σε σχέση με προηγούμενα θέματα που αναφέρθηκαν. Αν εξετάσουμε τώρα το θέμα της αρμοδιότητας και τις μεμονωμένες περιπτώσεις, διαπιστώνουμε ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα για την εφαρμογή των κανόνων. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει αρκετή διάσταση απόψεων προς το παρόν. Γι' αυτό και απαιτούνται περισσότερες συζητήσεις. Οι χώρες μέλη επισήμαναν το θέμα της απόσπασης, αλλά και το έργο του οργανισμού, των οργανισμών, των γραφείων προσωρινής απασχόλησης και να αποκλειστούν οι εργαζόμενοι ε, μέσω τέτοιων γραφείων προσωρινής απασχόλησης από το πεδίο εφαρμογής οδηγίε. Όπως όμως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πλειοψηφία των κρατών μελών θεωρεί ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι θα πρέπει να οριστούν με ακρίβεια και τα κράτη-μέλη να ορίσουν τους τομείς για τους οποίους ε, επιτρέπεται τέτοιου είδους εποχιακή απασχόληση. Εδώ υπάρχουν και εθνικές ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εποχής για να προσδιορίζεται η εποχιακή απασχόληση. Όπως είπε και ο κύριος Μωράης, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί κατάλληλη προστασία στους εργαζόμενους και να αποφευθούν περιπτώσεις εκμετάλλευσης ή κατάχρησης των διατάξεων. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η προστασία των διαταξεων εμας μας ενδιαφερει περισσότερη προστασια των εργαζομενων Και αν στο Συμβούλιο έχουμε το θέμα απόρριψη απόσυρσης και αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει να το εξετάσουμε γιατί αν ένας εργαζόμενος, ένας εργάτης δεν πλήρει τις προϋποθέσεις ε, για μια συγκεκριμένη δουλειά ή αν υπάρχουν προβλήματα κοινωνικής ασφάλισης ή φορολογίας ή με την ίδια την εργασιακή σύμβαση, όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να διευκρινιστούν. Πάντως στο Συμβούλιο σημειώθηκε πρόοδος ε, σε πολλά ζητήματα ουσίας και ευελπιστούμε ότι με βάση τα αποτέλεσματα αυτά θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και στην διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Τώρα έχουμε δύο ε, μέλη που θα απαντήσουν από ο κύριος Σκοφεράτη από την Επιτροπή Απασχόληση, η κυρία Παπαδοπούλου από την Επιτροπή των Γυναικών. Ο κύριος Σκοφεράτη πρώτα έχει το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Κλοντ Μωράης για τη συνεργασία αυτή. Εάν θέλουμε, όπως λέει η Κομισιόν, να ορίσουμε πολιτικές ε, για τη μετανάστευση που να είναι ομοιόμορφες χρειάζονται δύο πράγματα. Καταρχήν οι μεμονωμένες διατάξεις να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο, να ενταχθούν σε μια κοινή λογική. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία η οποία ευτυχώς υπάρχει μεταξύ της δικής σας Επιτροπής και της Επιτροπής Απασχόλησης. Στόχος ο οποίος είναι σαφής και τον συμμερίζονται όλοι. Ο στόχος λοιπόν είναι ε, αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να εργαστούν εύρυθμα, να μην υπάρχει ένα στοιχείο κινδύνου και να μπορέσουν ε, να εργαστούν κάτω από συνθήκες έτσι ώστε να μην επιβληθεί κοινωνικό dumping και να μην υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων. Να υπάρχει δηλαδή ένας ενιαίος κανόνας στην αγορά. Γι' αυτό όπως αναφέρθηκαν και ορισμένα στοιχεία, εγώ τα ε, αναφέρω, αναφέρομαι σε αυτά εντάχει, τα στοιχεία είναι τα εξή. Αν δεν θέλουμε να υπάρξει κοινωνικό dumping θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ίσες συνθήκες για τους ενδιαφερόμενους. Με αυτό θέλω να πω να υπάρχει ίση μεταχείριση για παρόμοια εργασία και έτσι θα μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το χάσμα στο οποίο βρίσκονται οι επιχειρήσεις μη χρησιμοποιώντας ε, εθνικούς ε, από την εθνική αγορά εργαζομένους, αλλά εργαζόμενους από τρεις χώρες, χωρίς να υπάρχει εξασφάλιση δικαιωμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση για να μην υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ και αθέμητος ανταγωνισμός. Όταν μιλάμε για μεταχείριση, θα πρέπει να αναφερθούμε στους, ε, στις συνθήκες συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή συλλογικές συμβάσεις έτσι ώστε να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για να έχουν αυτά τα πρόσωπα τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι άλλοι εργαζόμενοι. Δεν μιλάμε μόνο για τις, για τις συμβάσεις, μισθό, ωράριο, ασφάλεια, αλλά μιλάμε και για την ε, προσωρινή τους ε, κοινωνική θέση. Δηλαδή, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αξιοπρεπής εργασία, έτσι ώστε το πρόσωπο αυτό να μην υφίσταται αρνητικές ε, συνέπειες όπως η σε ένα συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο κοινωνικό ιστό και δαφικό ιστό. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παρατηρήσουμε, όπως φαίνεται και από την έκθεση του Κλοντ, να παρατηρήσουμε και να δούμε τι σημαίνει ίση μεταχείριση και ίσες συνθήκες. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αν λάβουμε υπόψη τις ηλικέ συνθήκες και τα δικαιώματα, μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να δούμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής και ο χρόνος εφαρμογής. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το εξής. Δεν θα πρέπει όλα να τα ορίσουμε ως εποχικές εργασίες, διότι πολλές φορές αυτό προσπάθησαν να κάνουν πολύ. Υπάρχει, ε, ας πούμε, προσωρινή εργασία, ευκαιριακή εργασία που δεν είναι εποχική. Άρα δεν θα πρέπει να επιβάλλεται ο εποχικός χαρακτήρας. Να δούμε τι πραγματικά είναι εποχική εργασία και όχι προσωρινή ας πούμε. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη μία ευρύτερη ερμηνεία από αυτή που ορίζουμε εμείς, διότι οι εποχές στην Ευρώπη δεν είναι ίδιες μεταξύ Βορρά και Νότου και στην ε, οργάνωση δεν έχουν τις ίδιες επιπτώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ευελιξία διαμέσου μιας συμφωνίας μεταξύ κοινωνικών εταίρων που να μην αλλοιώνει αυτές τις συνθήκες. Το τελευταίο θέμα αφορά το χρόνο, θέματα χρονισμού. Δηλαδή, μιλάμε ημερολογιακά όμως για τα απορροκυπευτικά ή για τις γεωργικές εργασίες λαμβάνουμε υπόψη το ηλιακό σύστημα και όχι το ημερολογιακό. Στον τουρισμό δεν ισχύει το ίδιο, δηλαδή ξέρουμε τι είναι ο καλακερινός τουρισμός και τι είναι ο χειμερινός ε, τουρισμός μέσα στα πλαίσια του, των 12 μηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και ελπίζω να Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και σε άλλους τομείς. Έχουμε και άλλους ομιλητές, λέει ο Πρόεδρος, γι' αυτό θα ήθελα να είσαστε ιδιαίτερα σύντομοι και να το λάβετε υπόψη, έτσι ώστε να αναφερθούν όλα τα ε, σημεία ε, το λόγο έχει η κυρία Παπαδοπούλου, εξ ονόματο τη Επιτροπή Γυναικών. Σύντομα. Στη σειρά μου να πω ότι ήμουν η συντάκτρια γνωμοδότηση από πλευρά τη Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητα των Φίλων προ την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η δική μα γνωμοδότηση έχει δει το θέμα από την οπτική γωνιά των γυναικών. Ε, γιατί σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Οικονομικής και του ΟΗΕ αλλά και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ένα σημαντικό ποσοστό εποχικών εργατών είναι γυναίκες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες, οι οποίες ε, μαστίζονται από τη φτώχεια, τον αναλφαβητισμό και ε, οπωσδήποτε από δύσκολε ηθίκες διαβίωσης και χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Αυτές οι γυναίκες όταν έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εργασία υπόκεινται σε αρκετές δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή τους και επιπρόσθετα αντιμετωπίζουν στερεότυπες αντιλήψεις περί φύλου, προκαταλήψεις, ε, ανισομιστία. Ε, διακρίσεις πολλές φορές δεν γνωρίζουν τα δικά τους δικαιώματα και οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν εκείνα τα μέτρα για να υπάρχει η δημιουργία ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος. Εμείς συμφωνούμε με την έκθεση που έχει κάνει ο κύριο Κλωτ Μωράες γιατί ακριβώς ο στόχος είναι να υπάρχουν ε, ξεκάθαροι όροι επαναπατρισμού των εποχιακά εργαζομένων και των γυναικών, να υπάρχει ευχαίρεια διασφάλισης του δικαιώματο ξανά επιστροφή στη χώρα όπου εργάζονται, να διασφαλίζεται η ίση αμοιβή και η διάρκεια παραμονή να είναι καθορισμένη. Και όσον αφορά ειδικά τι γυναίκε, έχουμε εισηγηθεί να υπάρχουν ακριβώ συστηματικοί έλεγχοι των καταλήμματων στα οποία διαμένουν, περιοδική έλεγχη και κυρώσει όταν οι εργοδότε δεν τηρούν αυστηρά συνθήκε αξιοπρεπού διαβίωση να διασφαλίζεται η προστασία τους όταν είναι έγκυοι ή όταν έχουν ε, προβλήματα υγείας και οπωσδήποτε να υπάρχουν εκείνοι μηχανισμοί καταγγελίας παραπώνων για εκμετάλλευση ή κακομεταχείριση. Θεωρώ ότι με τις δικές μας προτάσεις που εσωματώνονται και στην έκθεση του κ. Μωράες ε, έχουμε ενώπιον μας ένα, μια, κάποιες λύσεις για ένα πολύ ευαίσθητο και καυτό θέμα των ημερών. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο. Να παρέμβετε λοιπόν για 1,5 λεπτό. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μωράη, τον εισηγητή μας, για την εξαιρετική του εργασία και για την εκτενή και επικοδομητική παρουσίαση που έκαναμε στα πλαίσια της συνεργασίας για την ε, έκθεση αυτή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Ως προς τα θετικά σημεία της έκθεσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεχόμαστε την εξαμηνία διάρκεια της εποχικής εργασίας με βάση τους 12 μήνες και κατανοούμε, αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο εισηγητής για να ορίσει τους τομείς εποχικής εργασίας. Επίσης είναι θετικό το ότι αποτελεί ε, στέγη και ποια μέτρα, ποια ειδικά μέτρα ε, λαμβάνονται. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερες ρήτρες διασφάλειας σε σχέση με πληροφορίες τη στιγμή που δεν θα υπάρχει διοικητικός φόρτος που θα επιβραδύνει τη διαδικασία. Τέλος, θα ήθελα να θεωρήσω ευπρόσδεκτους τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου, καθώς και την επέκταση κυρώσεων κατά των εργοδοτών όταν υπάρχουν παρατυπίες. Τώρα θα ήθελα να σταθώ σε ζητήματα ζωτικότερης σημασίας για τη δική μας ομάδα και καταρχήν ορισμένες ε, επικρίσεις ή ορισμένα κρίσιμα σημεία. Θα ήθελα, όπως είπε και ο εισηγητής, να δούμε ποιες είναι οι μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με εκείνους οι οποίοι παράνομα διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τροπολογίες 6 και 18. Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα σχετίζεται με τον απότερο στόχο της οδηγίας. Η οδηγία αυτή αφορά τη νόμιμη μετανάστευση αυτό μας απασχολεί εξ αρχής. Κατανοώ αυτά, που, ε, αυτά στα οποία αναφέρεται ο εισηγητής, αλλά αυτά ε, βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής που αφορά την ε, κυκλική μετανάστευση επίσης. Δεν μας απασχολεί το θέμα των παράνομων μεταναστών, εκείνων που προσπαθούν παράνομα να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι φαίνεται ότι υπερτιμούμε τους παράνομους μετανάστες σε σχέση με αυτούς που νόμιμα θέλουν να μεταναστεύσουν. Βεβαίως υπάρχει εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων και θέλουμε να τους προστατεύσουμε, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν κυκλώματα που προσπαθούν να βρουν παραθυράκια και νέους τρόπους εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και νέες ε, μεθοδολογίες, δηλαδή λένε στους μετανάστες μπείτε παράνομα και μετά θα βρείτε το δρόμο σας. Αυτό γίνεται και με τη διαδικασία ασύλου. Οι συνάδελφοι ξέρουν ε, επακριβώς τι εννοώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επαναλαμβάνω λοιπόν, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθώ, μία, ένα από τα βασικά μας μελήματα εξ αρχής είναι να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κατάχρηση αυτής της οδηγίας, ιδιαίτερα με υπέρβαση διαμονής. Θα προσπαθήσουμε να το ξαναδούμε και με τροπολογίες και με συζητήσεις για να βελτιώσουμε το κείμενο και να μειώσουμε το, να μειώσουμε, να περιορίσουμε τον κίνδυνο υπέρβασης ε, της άδειας παραμονής. Επίσης, ένα ε, άλλο σημείο που είναι απότοκο του προηγούμενου είναι να μην υπάρχει κατάχρηση της οδηγίας. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε μία νέα οδηγία η οποία θα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να έχουμε θεωρητικές συζητήσεις και αποφάσεις οι οποίες δεν θα τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε ορισμένα ζωτική σημασία ζητήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να έχουμε καλά αποτελέσματα κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, υπάρχουν και άλλα σημεία, αλλά θα είμαι σε στενή συνεργασία με τον εισηγητή και θα τα προωθήσω εκεί. σας ευχαριστω Πέντε Πεντέμιση λεπτά, κύριε Παπα-Νικολάου μου. Σας ευχαριστώ για αυτά που λέτε, αλλά δεν θα προλάβουμε να συνεχίσουμε έτσι. Χρειάζεται και κάποια αυτοσυγκράτηση. Ε, παρακαλώ, υπόλοιποι Δύο λεπτά έκαστος. Εμείς δεν προλαβαίνουμε. Θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Έχουμε και άλλα θέματα στη μέση διάταξη. Ο κύριος Thank you, Chair. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το δίλεπτο. Καταρχάς, ε, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Κλοντ Μωράς. Είχα επανειλημμένες συναντήσεις μαζί του και έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε για να καταλήξει σε συμβασμό και για τις τροπολογίες νομίζω είναι στη σωστή κατεύθυνση. Καταρχήν η ομάδα των φιλελευθέρων είναι υπέρ ενός κανονισμού ε, για τη ρύθμιση ε, της λειτουργίας και αυτών των εργαζομένων. Είναι ένα βήμα προς τα στη σωστή κατεύθυνση για την ενιαία αγορά. Μερικά σχόλια. Ο εισηγητής προτείνει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, μια διετία για τους παράνομα διαμένονται στην Ένωση. Να το σκεφτούμε γενικά, δεν είμαι υπέρ αυτή της ρύθμισης ή να κάνουμε ειδικέ χάρες σε αυτούς που στο παρελθόν παρανόμησαν. Πρέπει να το σκεφτώ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα. Στην τροπολογία 20 κάνει μια πρόταση ο κύριος Μωράες. Η πρόταση με βρίσκει σύμφωνο στην αρχή, αλλά στο τέλος λέει ότι ε, θα αφορά τη γεωργία, τη φυτοκομία και τον τουρισμό, το είπε, και τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν την επέκταση της εφαρμογής επιπρόσθετες δραστηριότητες κουλουπού, κουλουπού, και στο τέλος λέει υπό τον όρο ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι χρήσιμοι και θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να ενέχονται. Αλλά η τελική συμφωνία για τους νόμους στα κράτη-μέλη μας είναι πάντα η Βουλή και όχι η κοινωνική εταίρη. Ε, αυτό θα πρέπει να εγκρίνουμε. Ο συμβασμός για τη στέγαση είναι καλός. Εντάξει, 100% δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα του εργοδότη που θα του στεγάσει να είναι μια κατάλληλη στέγη για όλου. Κατάλληλες συνθήκες για τον καθένα, όχι μόνο για τους εποχικούς εργαζομένους. Και πάλι είναι και θέμα της κυβέρνηση να τα φροντίζει αυτά. Και συμφωνώ με το σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ. Το σημαντικότερο με αυτή την νομοθεσία είναι ο έλεγχος, πώς θα ε, εφαρμόζεται και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε ε, το γεγονός ότι μόλις εγκρίνουμε αυτό τον κανονισμό ή την οδηγία ε, να ε, βεβαιωθούμε ότι θα εφαρμόζεται σωστά και να φεύγει ο κόσμος μετά το εξάμεινο που επιτρέπεται να είναι εδώ. Ευχαριστώ. Και δεν μετρήσατε και το χρόνο. Α, πώς δεν μετρήσατε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαρχεντίνη, η σειρά σας τώρα. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση ε, του Κλοντ Μωράης για τις τροπολογίες του είναι καλές, η πρόταση είναι καλή μάλλον, αλλά είναι πολύ μετριοπαθής. Καλό είναι να έχουμε οδηγία για τους ε, εποχικούς εργαζομένους, αλλά ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο με τη μετανάστευση για λόγους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ο κύριος Μωράες, ε, αλλά τουλάχιστον είναι η πρώτη ευκαιρία να συζητήσουμε για την νόμιμη μετανάστευση για εκείνους που δεν έχουν ε, τη μεγαλύτερη δυνατή μόρφωση και τα περισσότερα προσόντα. Έρχομαι μέσως στο θέμα των λαθρομεταναστών που ήδη διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο και η κίνηση να τους επιτρέψουμε να ε, ζητήσουν να ενταχθούν σε αυτό το θέμα. Βέβαια όταν εργάζεσαι έξι μήνες όλοι γνωρίζουν ποιος είσαι και πού βρίσκεσαι και θα σε αναγκάσουν να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτός δεν είναι τρόπος ε, τακτοποίησης και νομιμοποίησης παρανόμων μεταναστών. Τους δίνει την ευκαιρία να εργαστούν και ε, να φύγουν με ένα καλό ε, τρόπο ε, αξιοπρεπή, με ψηλά το κεφάλι, ε, να γυρνάει στην οικογένεια του ο καθένας και να δείξει ότι κάτι έκανε, ότι έβγαλε χρήματα, ότι είχε δουλειά και όχι ότι τον έχουν διώξει με απαγόρευση επανεισόδου. Υπάρχουν λοιπόν ήδη παράνομοι μετανάστες και ο βασικός στόχος όμως των πρασίνων σε αυτή την οδηγία είναι επιτέλους να δοθεί μια νόμιμη εναλλακτική λύση ε, σε κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό ή φυσικό σχεδόν παντού στην Ένωση. Οι παράνομοι μετανάστες εργάζονται ε, και πολύ συχνά σε πολύ σκληρές και δύσκολες συνθήκες. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, θα μπορούσε να βοηθήσει και δεν καταλαβαίνω τα κόμματα εκείνα που λένε ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι θα αυξήσουν, λέει, τη λαθρομετανάστευση. Γιατί θα παραμένουν όταν θα λύγει η άδειά τους. Αυτό αγνοεί, παραγνωρίζει την πραγματικότητα. Σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαίνει αυτό. Ήδη απασχολούνται λαθρομετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν ε, κανένα τρόπο μέχρι τώρα να τακτοποιήσουν, να νομιμοποιήσουν ε, την παρουσία τους. Αυτό είναι το κλειδί λοιπόν και είμαι πρόθυμη να δεχθώ έστω αυτό το ε, περιορισμένο χρονικό διάστημα του εξαμήνου και να περιορίσουμε και συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Θα κάνουμε και κάποιες τροπολογίες ε, για το καθεστώς των εποχικών εργαζομένων και τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ. Μέχρι τώρα έχουν, με έχουν μάθει οι συνάδελφοι και ξέρουν ότι είμαι υπέρμαχος του πακέτου για τη μετανάστευση. Και χαίρομαι που και στην περίπτωση αυτή έχουμε ως εισηγητή μας ε, τον Κλοντ Μωράες, γιατί και λογικός είναι και συνετός και ικανός ε, να προωθήσει τις συζητήσεις για το θέμα αυτό. Ναι, είμαι υπέρ της ρύθμισης της εποχιακής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους επικούς τρίτων χωρών, αλλά όπως και στο παρελθόν θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι και οι εποχικοί απασχολούμενοι ε, μάλλον η εποχιακή απασχόληση είναι μια απασχόληση και για τους ε, ενδοκινοτικούς, ε, γιατί και εκείνοι μετακινούνται και προσφέρουν εποχιακά εργασία σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσθέσουμε και τη δική τους θέση. Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές συνθήκες, τη στέγαση κτλ. πιστεύω ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές, οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται, μετακομίζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε υψηλότερες προσδιαγραφές για τους εξωκοινοτικούς από ό,τι για τους ενδοκοινοτικούς. Ε, πέραν τούτου θεωρώ ότι η πρόταση είναι σε καλή κατάσταση. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση. Θετικά, επιγραμματικά, ίση μεταχείριση, πολύ σημαντική και παίζει και σπουδαίο ρόλο. Εντάξει, είναι και στην έκθεση και θα πρέπει να κριθούμε και σε αυτό και σε άλλες εκθέσεις. Τι γίνεται με τους ε, εργαζόμενους που παραβιάζουν την ομοθεσία, εντάξει να το συζητήσουμε και πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε και για τις κυρώσεις. Έλεγχοι επιθεωρήσεις, πολύ ωραία, είμαστε και εδώ υπέρ, δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, να ενισχυθούν και αυτό που μου αρέσει πολύ είναι το θέμα της στέγασης. Ε, ε, αυτό το, το στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας το τονίζεται πολύ ωραία. Προβλήματα. Αίτηση ε, στο εσωτερικό των κρατών μελών και η διετία. Νομίζω ότι εδώ βοηθάμε να έρθει η παρανομία. Διότι ε, είναι γεγονό ότι ήδη εργάζονται οι παράνομοι μετανάστες, ακριβώς παράνομα, στη Μαύρη, σε πολλά κράτη-μέλη, ε, άτυπα. Και εκεί έχουμε ανοίξει τις για την πιο ικτρή εκμετάλλευση. Θα πρέπει να έχουμε συμφέρον να το καταργήσουμε αυτό. Και δεν το καταργούμε εάν αφήνουμε εκτός αυτούς τους εργαζομένους, οι οποίοι ήδη εργάζονται, θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να νομιμοποιήσουν την κατάσταση και την παρουσία τους και να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ρυθμούς που αποφασίζουμε και με τα μεταβατικά κτλ. στην οδηγία. Να το σκεφτούμε παρακαλώ σοβαρά αυτό. Και είμαι και στη διάθεσή σα να συζητήσω αν θέλετε και τη διετία, μήπως μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο. Αλλά επί της αρχής συμφωνώ και το θεωρώ πολύ σημαντικό οι ορισμοί, τι εστί εποχική απασχόληση, δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει και εγώ που το παραδέχομαι. Έγινε μια απόπειρα ορισμού με τους διάφορους κλάδους. Εντάξει, λογικό μου φαίνεται αυτό, αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο. Και ένα τελευταίο. Θα ήθελα πιο σαφή διατύπωση για τα δικαιώματα των εποχικών εργαζομένων και αυτό να το ξαναδούμε κάπου χωριστά σε μια ειδική παράγραφο να ορίσουμε τι δικαιώματα έχουμε γιατί αυτό δεν έχει καλυφθεί επαρκώς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έντσιου. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, κλώτη για την έκθεση που συνέτεξε, γιατί προτείνει να καλύψει τα χάσματα που υπάρχουν και μιλάει για βελτίωση σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας. Θα ήθελα να ε, στραφώ μόνο στις ε, κυρώσεις που ισχύουν για τους εργοδότες αν δεν τηρούν τη νομοθεσία γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εποχικοί μπορούν να δουλεύουν σε συνθήκες ημισκλαβιάς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο κυρώσεων και να μιλήσουμε και για τους μεσάζοντες και για τους οργανισμούς τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, διότι αυτοί οι οργανισμοί είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με τους ενδυνάμει εποχικούς και θα πρέπει να τους ενημερώνουν σε σχέση με τα δικαιώματά τους μέσα στα πλαίσια διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Μωράης να προσπαθήσετε να ενσωματώσετε όλα αυτά τα στοιχεία που ακούσατε και από τις Επιτροπές Απασχόλησης και Γυναικών, δηλαδή των ε, κυρίων Κοφεράτη και Παπαδοπούλου. Έχετε το λόγο κύριε Μωράης. Ευχαριστώ. Γνωρίζω κι εγώ ότι έχουμε καθυστερήσει, αλλά επειδή τιμώ τους ε, Σκιώδης και τους ε, Κοφεράτη και Παπαδοπούλου. Βεβαίως όλοι ε, έχουν ασχοληθεί με την έκθεση. Είναι σαφές ότι την έχουν διαβάσει και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια πραγματική συζήτηση πέρα από την τομεακή προσέγγιση ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ανεργία, έχουμε λιτότητα. Το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα πολύ σκληρό θέμα και ζωτική σημασία. Θα πρέπει να αποφύγουμε την εκμετάλλευση των ανθρώπων και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους αποχικούς και για τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Θα ήθελα λοιπόν να στραφώ στο θέμα του κυρίου Μούλντερ για τους κοινωνικούς εταίρους μίλησε για κάτι το πολύ σαφές και αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνουν σαφείς ε, ε, συζητήσεις στον τομέα των κατασκευών. Τον απέκλεισε αυτό το τομέα διότι δεν έχει εποχικό χαρακτήρα. Εάν ένα κράτος μέλος το αποφασίσει τότε έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αλλά οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συμβουλεύσουν αλλά σε τελευταία ανάλυση τα κράτη-μέλη ελέγχουν την κατάσταση. Αυτό είναι απόλυτα σαφές και ανακύπτει κάθε φορά από τις συζητήσεις. Ο κύριος Παπανικολάου ήταν απόλυτα σαφής για το τι, τον βρίσκει σύμφωνο και τι όχι. Ξέρω, ξέρω με τι να έχω να κάνω. Ε, ως προς τα δύο σημεία που δεν τον βρίσκουν σύμφωνο είναι πολύ περίπλοκα. Το ένα ίσως λιγότερο από το άλλο. Το ένα ε, αφορά την υπέρβαση ε, διαμονής Ποιο είναι δηλαδή παράνομος και ποιο όχι. Μπορούμε να το συζητήσουμε πίνοντας τον καφέ μας. Το άλλο είναι ε, ένα πρακτικό ζήτημα, γι' αυτό προσπαθώ να γεφυρώσω το χάσμα, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια αποσαφήνιση. Ο Γιάν Μόλτερ είναι πάντα ε, απόλυτα σαφής για το τι του αρέσει και τι όχι. Άρα έχω μια πολύ καλή βάση εργασίας και τι μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω. Σαρτζεντίνη και Έρνστ. Ίσως ε, κινούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ίσως είμαι ιδιαίτερα ε, μετριοπαθής ως προς την γεφύρωση, αυτό το γεφύρωμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Βέμπερ λέει ότι είμαι πολύ λογικός, αλλά μπορώ και να μην είμαι αν δεν με θέλετε. Εξαρτάται από το τι θέλετε. Ξέρετε ότι μπορώ, ξέρετε ότι μπορώ να είμαι και το αντίθετο. Α, όχι, η κυρία Λάντφορτ το ξέρει. Το ξέρει ακόμα καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθείτε να πείτε και το εκτιμώ ιδιαίτερα είναι ότι ε, αυτές ε, οι παράμετροι είναι πολύ σημαντικοί. Αυτό αφορά και την απόσπαση και τους εποχικούς. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα πώς το προσεγγίζουν οι σκιώδεις, διότι είναι ιδιαίτερα ειλικρινείς και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για να έχουμε μια πραγματική συζήτηση και να κάνουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, όπως είπε και ο κύριος ε, Κοφεράτη, με βάση τον απότερο στόχο μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά να αλλάξουμε τις συνθήκες, να αλλάξουμε έναν τομέα. Θα είναι πολύ δύσκολο βεβαίως, αλλά εύχομαι να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Απασχόλησης έτσι ώστε σε κάποιο στάδιο να έχουμε μια ισορροπημένη ε, οδηγία που θα υποστηρίξουν όλοι. Ευχαριστούμε Κλοντ. Και ευχαριστώ όλους και για τη συζήτηση. Ήταν πολύ χρήσιμη και νομίζω ότι βάλαμε τα θεμέλια της συζήτησης και μπορούμε να ορίσουμε την προθεσμία για την κατάσταση των υπολογιών στις 12 Ιουλίου το μεσημέρι μια ναι, και η Επιτροπή Απασχόλησης έχει ορίσει η διορία για τις τροπολογίες την 22 Ιουνίου. 22 Ιουνίου για την Επιτροπή Απασχόληση το μεσημέρι και εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη 12η Ιουλίου 12 το μεσημέρι επίσης. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι συναφές με το προηγούμενο, με τα δύο προηγούμενα, τα 20 και 21, γιατί και το 22 αφορά το πακέτο της μετανάστευσης. Διαδικασία ενίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας. Και αυτή η πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα, μια συνιστόσα του πακέτου μετανάστευσης. Η εισηγήτριά μας θα μας ενημερώσει για την πορεία των συζητήσεων σε ό,τι αφορά την οδηγία που προβλέπει διαδικασία ενία αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας υπηκοτρή της χώρας για εργασία και παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μάρτιο 24 του μηνός το Κοινοβούλιο ψήφισε. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ματιέ και θα μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα στον πρώτο τριμερή διάλογο της 23ης του μηνός, ώστε να καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε την υπόθεση αυτή στη δεύτερη ανάγνωση. Κυρία Βερονίκ Ματιέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως μας είπε ο Πρόεδρος, στις 23 Μαρτίου καταλήξαμε σε συμφωνία μετά την υιοθέτηση της έκθεσης για τη διαδικασία ενιαίας αίτησης και συνεχίσαμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Στις 23 Μαΐου έλαβε χώρα ο πρώτος τριμερής διάλογος όπου καταφέραμε να διευκρινίσουμε τη θέση μας απέναντι στο Συμβούλιο. Και μάλιστα ε, ε επιβεβαιώθηκαν τα 107 σημεία του Κοινοβουλίου, αλλά έχουν απομείνει κάποια επίμαχα σημεία που είναι σημεία τριβής και μας παρουσίασε το Συμβούλιο στον τριμερή διάλογο. Το πρώτο αφορά την αναφορά στους πίνακες αντιστοιχία. Όπως ξέρετε, πρόκειται για ένα οριζόντιο θέμα που απασχολεί μια διοργανική ομάδα εργασίας. Δεν θα αποφαθώ καθόλου για το θέμα αυτό. Το δεύτερο σημείο αφορά την μέγιστη προθεσμία για τη χορήγηση αυτή τη ενιαία αίτηση. Στην Ολομέλεια ψηφίσαμε το τρίμηνο. Το Συμβούλιο προτιμά τέσσερι μήνε και ίσω αυτό το θέμα εξεταστεί στι τελικέ διαπραγματεύσει. Μάλιστα, στην Ολομέλεια είχαμε ονομαστική ψηφοφορία και το εγκρίναμε με 584 ψήφου υπέρ. Τρίτο θέμα. Οι συμπληρωματικέ πληροφορίε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι και το σημείο αυτό το εγκρίναμε με 584 ψήφους υπέρ, με ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Και είναι το μόνο σημείο στο Συμβούλιο που υπόκειται στην ανασχετική μειοψηφία. Γιατί πολλές χώρες θέλουν να, ε, η ενιαία αίτηση να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες επιπρόσθετες ε, για τον εργαζόμενο. Μετά τις διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο μας κοινοποίησε μια συμβαστική πρόταση. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική αυτή πρόταση, προβλέπει οι πληροφορίες να είναι ίδιες με αυτές που περιλαμβάνονται σήμερα στην άδεια εργασίας, δηλαδή ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, τόπος, είδος απασχόλησης και αμοιβή. Επιπλέον, η μία των πληροφοριών αυτών είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι μπορούμε, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη και πολλών ασκιωδών εισηγητών, Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση του Συμβουλίου γιατί είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να καταπολεμήσουμε τη λαθροεργασία και την εκμετάλλευση εργαζομένων τρίτων χωρών. Είναι ισορροπημένη αυτή η συμβαστική πρόταση. Μια και ο κατάλογο των πληροφοριών είναι εξαντλητικό και όχι ενδεικτικό, δεν υπόκειται δηλαδή στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τον τύπο, το format το είδο ε, αίτηση που θα χρησιμοποιείται για την ενιαία αίτηση δεν περιλαμβάνει την συμπεριλήψη ορισμένων πληροφοριών ε, σε, λόγω έκταση και αυτό μπορεί να συμπεριληφθούν σε, ένα, σε ηλεκτρονικό ντοσιέ ή σε έγγραφο. Βέβαια, έτσι θα μειωθεί το κόστο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και για τη δημόσια διοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο προτείνει μία, μία ξεχωριστή παράγραφο για την ισότητα μεταχείριση ό,τι αφορά τις υπηρεσίες απασχόλησης. Συμφωνούμε γιατί έτσι δεν θα περιορίσουμε την πρόσβαση αυτή και θα επιτρέψουμε στους ανέργους που είναι αυτοί που το χρειάζεται περισσότερο να έχουν πρόσβαση. Και εδώ το Συμβούλιο είναι πιο γενναιόδωρο από αυτό που ψήφισε το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια. Πέμπτον, ισότητα μεταχείρισης σε ό,τι αφορά πρόσβαση στην παιδεία και την επαγγελματική κατάρτιση. Το ψηφίσαμε και αυτό στην Ολομέλεια με 463 ψήφους υπέρ σε ονομαστική κλίση, ονομαστική ψηφοφορία το Συμβούλιο περιόρισε την ίση μεταχείριση σε αυτούς που πραγματικά εργάζονται. Εμείς ε, ζητήσαμε να περιληφθούν και οι άνεργοι. Έκτον, σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των συντάξεων, το Συμβούλιο θέλει να συναρτήσει αυτή την εξαγωγή των συντάξεων με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας. Εμείς ε, το θεωρήσαμε ως ε, νευραλγικό σημείο Είμαστε υπέρ της μεταχείρισης και περιμένουμε να μας προσεγγίσει περισσότερο το Συμβούλιο στο θέμα αυτό, να συγκλίνει περισσότερο μαζί μας. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Υπάρχουν και άλλα πιο τεχνικής φύσης, μάλλον γλωσσικής. Θα τα διευθετήσουμε και αυτά, αλλά Χωρί ιδιαίτερες δυσκολίε. Μετά τον τριμερή διάλογο οργανώσαμε συνεδρίαση των σκιωδών την προηγούμενη Τρίτη στο Στρασβούργο και καταφέραμε να καταλήξουμε στην εξή συμφωνία που θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο. Δεχόμαστε τη συμβαστική πρόταση του Συμβουλίου για τα άρθρα που αφορούν τις συμπληρωματικέ πληροφορίε και την τετράμινη διάρκεια για την ε, επεξεργασία της αίτησης, αλλά ε, σε ό,τι φορά την ε, πρόσβαση και στις πληροφορίες ε, μένουμε στη δική μας στάση. Έχουμε τριμερή διάλογο και την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο στα πλαίσια της ε, δεύτερης ανάγνωσης. Ευχαριστώ τους και ηγητές που ήταν πολύ διαλλακτικοί και συνεργάσιμοι και είμαι έτοιμη να απαντήσω στις απορίες σας. Thank you, Ευχαριστώ, Βερονίκ. Θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για πάρα πολύ σύντομες παρεμβάσεις, αν θέλουν να μιλήσουν. Αλλά δεν θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην ημερησία διάταξη και πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και απλώ ενημερωνόμαστε για την κατάσταση των πραγμάτων. Από πλευράς Συμβουλίου, κυρία Βαλάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την κυρία Βατιού, την εισηγήτρια, για τις προσπάθειές της. Και εξ ονόματος του Συμβουλίου Θέλω να ευχαριστήσω και τις προηγούμενες προεδρίες, γιατί ξέρετε ότι αυτή η διαδικασία έχει προϊστορία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η οδηγία και μετά από μακρές διαπραγματεύσεις έχουμε την αίσθηση ότι δεν απέχουν και πάρα πολύ οι θέσεις ε, του Κοινοβουλίου από τη θέση του Βουλίου. Υπάρχει χώρος λοιπόν και ευκαιρία για συνεννόηση και για συμβιβασμούς. Όπως τόνισε ήδη η κυρία Ματιώ παραμένει σε εκκρεμότητα ένα πολύ σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, την ε, συγκροματική ενημέρωση, το Συμβούλιο Αποδεί πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα θέματα Και είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται ε, για τις εργασιακές σχέσεις ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, και για τη χορήγηση της άδεια εργασίας. Στο μέλλον ε, θα είναι ενιαία. Αλλά αν κάποιος θέλει επιπλέον πληροφόρηση, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει καθυστέρηση στη χορήγηση της άδεια. Και βεβαίω θα πρέπει πάντα να ισχύει αρχή της μεταχείρισης. Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί, να δείξει ευελιξία και να προσεγγίσει το θέμα από τη σκοπιά της ίσης μεταχείρισης. Παραμένουν και άλλα θέματα σε εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και την ενημέρωση των εργαζομένων, στην γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο ε, θεωρεί σημαντικό να διευκρινιστεί περαιτέρω αυτή η υπόθεση. Αυτό θα μπορούσε να το δεχτεί το Συμβούλιο. Και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, ε, τα συνταξιωτικά, ελπίζω να δώσει λύση ο τριμερής διάλογος ε, την άλλη εβδομάδα. Γιατί έχει ήδη προγραμματιστεί για την άλλη εβδομάδα. Και θα δώσει περισσότερες διευκρινήσεις, θα συμπληρώσει ε, το κείμενο. Σας λέω δεν απέχουμε πολύ σκέψη μας και στον τριμερή διάλογο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, uh, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμμερίζεται ε, τα θετικά σχόλια και της συζητήτριας και ε, του Συμβουλίου. Ε, νομίζουμε ότι θα βρεθεί ε, πλέον λύση νωρί τη δεύτερη ανάγνωση μετά από τέσσερα χρόνια διαβουλεύσεων. Ε, παραμένουν πολύ λίγα θέματα ε, και στα περισσότερα έχουν βρεθεί συμβιβασμοί. Συγγνώμη. Και τι γίνεται με τα στοιχεία που δεν χωράνε στην εναρμονισμένη άδεια εργασίας. Δεν ξέρω αν θα είναι με τρόπο ηλεκτρονικό ή άλλο, αλλά αυτό μπορεί να λυθεί. Για τις συντάξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ε, και σε αυτό το θέμα να μπορούν να μεταφέρουν τα συνταξιδευτικά τους δικαιώματα εργαζόμενοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα ίσονος σημασία εντό εισαγωγικών θέματα που εκκρεμούν ακόμα, όπως είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση των εργαζομένων, μπορούν να λυθούν την άλλη εβδομάδα στον τριμερή διάλογο και ε, παραμένει δεσμευμένη και προσιλωμένη προς την κατεύθυνση εξέβρισης λύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης εκφράζει την ελπίδα της να ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος μετά από τόσες συζητήσεις, παλινοδίες και αμφισβήτηση και να συμπληρώσει το πακέτο για τη νόμιμη μετανάστευση. Ε, πρόεδρος, είπαμε δεν θα γίνει συζήτηση, δεν θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Επιβεβαιώνουμε την εντολή της κυρίας Ματιού και της ευχόμαστε καλή τύχη για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Και θα θέλαμε να περάσουμε αμέσως στο επόμενο και τελευταίο για σήμερα το πρωί θέμα, χρησιμοποίηση των προσωπικών στοιχείων επιβατών, PNR. πρόταση οδηγίας για τη χρήση προσωπικών στοιχείων επιβατών για την ανείχνευση, πρόληψη, δίωξη και πάταξη ε, τρομοκρατίας. Είναι νέα πρόταση μετά την πρόταση του 2007. Αυτή η νέα πρόταση ε, αλλάζει σημαντικά δεδομένα. Θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή μας για το θέμα αυτό και μετά την Επιτροπή και το Συμβούλιο και στο τέλος θα κάνουμε μια μικρή ανταλλαγή απόψεων και θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε στις 12.30. Το λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Κύρκο. Μάλλον αδύνατο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Θα έλεγα να προβλέψουμε μόνο ένα τέταρτο για τη συζήτηση. Είναι απαράδεκτο τουλάχιστον για μένα ως ηγητή. Αυτό που σκοπεύω να κάνω και θα ζητήσω την βοήθεια της γραμματείας είναι να υποβάλω κάποια εισαγωγικά σχόλια και μάλιστα έχουμε εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής που ήρθαν επί τούτου για το θέμα αυτό και περιμένω εδώ και ώρα να τους ακούσουμε και προτείνω να ξαναβάλουμε το θέμα στην ημερή σε διάταξη ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό μεταξύ μας γιατί πραγματικά είμαι πολύ δυσαρεστημένος σε αυτή την κατάσταση είναι απαράδεκτη. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή γιατί είναι σημαντικό να αναλύσουμε διάφορες παραμέτρους στο στάδιο αυτό, γιατί ο συγγετής έχω λάβει πολύ υλικό, εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον, το ζήτημα επαναλαμβάνω είναι εξαιρετικά σημαντικό και μαζί με τους σκιώδεις συγγητές ήδη συναντηθήκαμε για να εξετάσουμε τα βασικά στοιχεία του θέματος αυτού και φαίνεται ότι πολλές, πολλά μέλη της Επιτροπής που ασχολούνται με θέματα PNR ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για την έκθεση. Θα είναι ένας ε, συναρπαστικός, μια συναρπαστική ευκαιρία για να εργαστούμε ζωηρά, επικοδομητικά και πολύ χρήσιμα. Από την μέχρι στιγμής πορεία μας ε, στα θέματα PNR μπορούμε ε, να αντλήσουμε πολλά συμπεράσματα από την προεργασία που έχει γίνει σε αντίστοιχε συμφωνίε με Καναδά, Αυστραλία και Ηνωμένε Πολιτείε. Πριν όμω ε, αρχίσω πολύ να ετοιμάζουν τι επιθέσει του ήδη από την αρχή, θα ήθελα να πω ότι παρόλο που πρόκειται για συμφωνία PNR, ουσιαστικά πρόκειται για μια ευρωπαϊκή συμφωνία PNR. Πιστεύω ότι παρά τι ε, βασικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε από πολλές απόψεις είναι μια συμφωνία διαφορετική και θα είμαι πολύ, προσεκτικό, θα είμαι πολύ προσεκτικός και στην προετοιμασία της έκθεσης για να φανεί αυτή η διαφορά και να τονιστεί ιδιαίτερα. Βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Είναι ενδιαφέρον ε, παρεμπιπτόντως ότι παρόλο που βρισκόμαστε στην αρχική φάση Τη διαδικασία και το μόνο έγγραφο που έχουμε μέχρι στιγμή στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχω λάβει γνωμοδοτήσεις σχεδόν από όλο τον κόσμο επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι και ευχαριστώ θερμά αυτούς που μου έστειλαν τις γνωμοδοτήσεις τους. Θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία και δείχνουν βέβαια ζωηρό ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρουσε αυτέ οι γνωμοδοτήσει. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις ως προς τη δική μου έκθεση. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί ο καθένας έχει σχολιάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν ενδιαφέρον αυτά τα σχόλια και τα διαβάζω, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι και οι σκέψεις για τη δική μου έκθεση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. έλαβα υπόψη και την γνωμοδότηση αυτή. Έχουμε το Συμβούλιο, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Είχαμε ε, επισυνημένη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τη μελέτη επιπτώσεων, το συνεπειών δηλαδή της πρότασης. Και μάλιστα ακόμη και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ζήτησε να γνωμοδοτήσει. Και μάλιστα συμφωνήσαμε η δική τους έκθεση να ακολουθήσει και να τη λάβουμε και εμείς πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Βέβαια το κυρίως θέμα της έκθεσης που σχετίζεται και με τις προηγούμενες εκθέσεις PNR, ε, συμφωνίες ε, PNR, αφορά το θέμα της διαχείρισης, επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, της χρήσης τους. Πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με θέματα δεδομένων. Ο κύριος Άλμπρεχτ, για παράδειγμα, γνωρίζουμε πόσο σημαντικά, είναι, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα. Το θέμα της ε, περίοδου φύλαξης, η χρήση τους, το κεντρικό σύστημα ή το αποκεντρωμένο σύστημα, ποιο είναι προτιμότερο. Όλα αυτά θα συζητηθούν. Είναι, θα είναι στοχευμένες οι πτήσεις, ε, κινδύνου, υψηλού κινδύνου ή θα καλύψουμε όλες τις πτήσεις, 100% δηλαδή συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων. Και κάποια άλλα θέματα που επισημαίνονται στην έκθεση του, στη γνωμοδότηση της, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θέματα διακρίσεων ή του profiling. Σε περίπτωση που δεν ε, επιλέξουμε την ε, πλήρη κάλυψη όλων των πτήσεων Και υπάρχει το θέμα των πόρων. Κόστος. Κάποιος θα πρέπει να πληρώσει ε, το λογαριασμό για όλα αυτά. Και εντάξει, πολύ εύκολα να την προτάσεις και όπως στο παιχνίδι με τις ε, μουσικές καρέκλες, όταν σταματάει η μουσική κάποιος θα πρέπει να αναλάβει, να, να, φανεί και να αναλάβει την ευθύνη. Θα πρέπει κάποιος λοιπόν να πληρώσει. Χθες μιλήσαμε για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση κατάχρησης ε, των, ή κακής χρήσης των δεδομένων. Επίσης το θέμα της επισκόπησης. Και αυτό το θέμα ενδιαφέρει. Χρειαζόμαστε έναν επιπλέον εποπτικό οργανισμό για την πλήρη επισκόπηση, την πλήρη επιτήρηση της διαδικασίας. Είναι όντως αναγκαίος ένας τέτοιος οργανισμός. Εξαρτάται από το πόσο κεντρικό θα είναι το σύστημα. Αναφέρθηκα ήδη στο profiling. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, δεν έχω καμία αφιβολία ότι το θέμα είναι σπουδαίο το είπα και στα αρχικά μου σχόλια που ήταν πιο οργισμένα, είναι αναμφίβολο ότι το θέμα είναι εξαιρετική σημασία και εξετάζοντα και την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και άλλε μα προτάσει σε προηγούμενε συμφωνίε PNR, γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε μια ισορροπία και ότι είναι χρήσιμη μια τέτοια συμφωνία για να αντιμετωπίσει τρομοκρατία και σοβαρά εγκλήματα, αλλά θα πρέπει και πάλι να είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει αυτή η πρόταση να χρησιμοποιείται ευρέω και πέραν των απαιτήσεων του Συμβουλίου και άλλων ότι πραγματικά θα χρησιμοποιηθεί για να ανεχρευθούν και να καταπολεμηθούν ε, εγκλήματα σοβαρά ή τρομοκρατικέ ενέργειε. Προσοχή λοιπόν να βρούμε αυτή την ισορροπία. Έχουμε κοινού στόχου. Πολύ σημαντικό το θέμα και πολύ σημαντικό να του υλοποιήσουμε. Είμαι υπέρ ε, ενός πνεύματος συνεργασίας και συλλογικού τρόπου ε, για την επεξεργασία της έκθεσης. Καλή θέληση υπάρχει. Θα είμαστε, καλό θα ήταν λοιπόν να ήμασταν επικοδομητικοί και συνεργάσιμοι. Θα γίνεται τακτική ενημέρωση, αλλά μην ξεχνούμε ότι υπάρχει το σημαντικό θέμα της ασφάλειας εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, Το έγγραφο εργασία θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο. Είναι αρκετά χρονοβόρη η διαδικασία. Από τη στιγμή που θα καταρτιστεί το έγγραφο εργασία, τότε νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε τη διεξοδική του ανάλυση, να προσθέτουμε, να αφαιρούμε, να συλλέξουμε και άλλες γνώμες και να καταλήξουμε σε μία εύχριστη, πρακτική και συνετή ορθολογική λύση, έχοντας διδαχθεί και από τις προηγούμενες μας συζητήσεις για άλλες συμφωνίες PNR. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί τελικά, θα έχουμε αίσιο αποτέλεσμα. Ίσως σήμερα μπορούμε να ακούσουμε κάποια προκαταρκτικά σχόλια, αλλά θέλουμε παρακαλώ την Γραμματεία να ξαναβάλει αυτό το θέμα στην σε διάταξη για να έχουμε νέα ευκαιρία για τη συζήτηση και μάλιστα σχετικά σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους για δύο λεπτά τον καθένα. Έχω εδώ την κυρία Νιτβέλτ την κυρία Λάτσφορτ, τον κύριο Αλφρέχτ και τον κύριο Φως. Και κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών και μετά Επιτροπή και το Συμβούλιο αν θέλουν. Η κυρία Νιτβέλτ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ε, συμφωνώ με τον εισηγητή ε, ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε σοβαρά και με την ησυχία μας. Οπότε καλά θα κάναμε να αναβάλουμε τη συζήτηση κανονική και να τη κάνουμε αργότερα, γιατί δεν μας επιτρέπει ο χρόνος τώρα να μπούμε σε βάθος και να κάνουμε έτσι επεστατωμένη ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να πω μόνο ότι χαίρομαι ε, που εργαζόμαστε με αυτή την ομάδα που αναφέρατε τη ομάδα PNR, αυτή την οικογένεια, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Ε, είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για όλα τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες, αλλά πάντα επαναλαμβάνω το ίδιο. Ε, τι είναι εδώ κομβικό και σημαντικό να αποδείξουμε και την αναγκαιότητα και την... Ε, αναλογικότητα. Και όσο περισσότερο εμβαθαίνουμε, τόσο πιο ε, βαθιά και εμπεριστατωμένη θα πρέπει να είναι η αιτιολόγηση και η δικαιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση αυτών των στοιχείων για τους στόχους που επικαλούνται. Ε, αρχίσαμε με αυτή τη συζήτηση, έγινε στο Στρασβούργο η αρχή την περασμένη εβδομάδα. Πάντως θα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να αποδείξουμε την αναγκαιότητα, γιατί όλες οι γνώμες που ακούμε αυτό τονίζουν ότι μέχρι τώρα η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής. Ευχαριστώ, η κυρία Λάτσφορτ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι στη συνήθεια ομάδα PNR. Είμαι ένα πνευματική στον πάγκο. Αλλά ενδιαφέρομαι πολύ για την πρόταση αυτή. Έχω παρακολουθήσει όλη αυτή τη συζήτηση πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και πιστεύω Ε, ε, είπαμε στον Ευρωπαίο Επόπτη προσωπικών δεδομένων πόσο σημαντική είναι η δουλειά του και πόσο χρήσιμη και η γνωμοδότηση και για αυτή την υπόθεση PNR και πρέπει να σας πω ότι είναι πραγματικά ε, εξοντοτική η γνωμοδότηση, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο κριτήριο της αναγκαιότητας ούτε της αναλογικότητας και ε, κάνει και ένα παραλληλισμό πολύ ενδιαφέροντα με την οδηγία για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εναρμόνιση, δεν υπάρχει και ασφάλεια δικαίου στα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνετε ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Ε, και υπονομεύεται έτσι η διάταξη περί περιορισμού των σκοπών ή των στόχων. Το ίδιο ισχύει και στη διατήρηση προσωπικών στοιχείων. Και θα πρέπει μόνο αναπερίπτωση να χρησιμοποιούνται και όχι μαζικά. Πολύ ειλικρινής και αν δεν ήταν τόσο ευγενής ο ίδιος θα ήταν αυτό πολύ απότομο και βίο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλητικό ενδεχομένω υπάρχουν κάποιες ε, στατιστικές μη διαφοροποιημένες ε, σχετικά με τα εγκλήματα που συνδέονται με ναρκωτικά και είναι σαν να δικαιολογούν έτσι όλα τα λαθρεμπόριο, την ε, χρήση ναρκωτικών, την κατοχή. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. στη μελέτη αντικτύπου λέει και αναφέρεται στο Βέλγιο 95% όλων των συλλήψεων για τα ναρκωτικά βασίζονται στο PNR. Το Βέλγιο όμω δεν έχει καν ένα σύστημα που να συλλέγει συστηματικά στοιχεία τέτοια ε, καταστάσεων επιβατών. Δεν ξέρω, θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ σοβαρή και βαθιά ανάλυση αυτής της πρότασης, διότι δεν είναι πολύ καλά εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη. Ευχαριστώ. Κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κέρχοπ για την εισαγωγή του έκανε σημαντικά σχόλια και παρατηρήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε και θα συνεργαστούμε καλά. Και πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Σε τόση συντομία δεν μπορούμε να το διεκπαιρεωσουμε αρων αρων Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε και άλλη συνεδριάση εδώ στην Επιτροπή για αυτό το θέμα. Τώρα πάρα πολύ σύντομα εγώ να σας πω ότι για τα θέματα αρχής τα είπε και η Σάρα Λάτφορτ μόλις Έχουμε τη γνωμοδότηση και ε, του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων, αλλά και νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου, επί παραδείγματι, λένε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και ε, ως προς τη συνταγματικότητά του και ως προς το κατά πόσο τηρεί το χάρτη των Θεμελιδών δικαιωμάτων. Εχθές ε, μιλήσαμε για τη διατήρηση στοιχείων ε, τηλεπικοινωνιών. Είναι πράγματα πάρα πολύ γνωστά και συμφωνεί η Επιτροπή μας ότι θα πρέπει να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της οδηγίας και θα τα βρούμε μπροστά μας και στο PNA και στη διατήρηση στοιχείων επιβατών. Και θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη η επιβεβλημένη διατήρηση στοιχείων και ε, συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, ε, αναπερίπτωση. Ε, αυτό γίνεται ήδη από σήμερα σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες. Εάν κάποιες αστυνομικές αρχές έχουν μια υποψία, μπορούν ήδη από σήμερα να κοιτάξουν τα στοιχεία του επιβάτη και να δουν από πού έκανε την κράτηση του εισιτηρίου κτλ. Αλλά το θέμα στην οργανωμένη εγκληματικότητα και στην τρομοκρατία προσπαθούν να αναγνωρίσουν κάποιες προπαρασκευαστικές δράσεις και συμπεριφορές. Αυτό θα πρέπει να συνδέεται με πρόσωπα, με συγκεκριμένους επιβάτες. Δεν μπορεί να γίνει με στατιστικές, με αξιολόγηση, αξιοποίηση, επεξεργασία στοιχείων, με έρευνες, ανακρίσεις των διοκτικών αρχών. Πρέπει οπωσδήποτε να συνδέονται με πρόσωπα. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα ε, και απέναντι της πολίτες μας, αλλά και νομικό και της ένομης τάξης. Ευχαριστώ, κύριος Φως. Ευχαριστώ, Ίγκα. Καταρχάς, θα ήθελα να υποστηρίξω και πάλι αυτό που είπε ο Τίμωθη. Σε αυτό το σύντομο διάστημα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και όντως χρειάζεται χρόνος. Ε, αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο Και το είδαμε και στο παρελθόν. Αλλά εξακολουθεί να με απασχολεί. Υπάρχει κανένα αντικειμενικό επιχείρημα για αποκεντρωμένο σύστημα PNR. Τι εννοώ. Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει να έχουμε ένα σύστημα κεντρικά κάπου. Το αποκεντρωμένο μπορεί να το κάνει από μόνο του το κάθε κράτος ξεχωριστά. Γιατί να έχουμε οδηγία η ευρωπαϊκή πρόταση. Για μένα η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι μόνο εφόσον υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα και για το κόστος. Και ε, υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι το κεντρό μένο σύστημα κοστίζει 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κεντρικό 87. Μήπως να το ξανασυζητήσουμε, ε, αν υπάρχει ε, σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία να είναι κεντρικό αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Φως. Ο κύριος εσύ ήθελε το λόγο. Εντάχει, θα ήθελα να πω ότι ο Σκιώδης δεν μπόρεσε να έρθει εδώ, αλλά συμφωνώ με τη μεθοδολογία που εισήγαγε ο κύριος Κέρκοπ, καθώς και αυτά που ε, είπε στις γενικές γραμμές και θα τα στην Κάρμεν Ρομέρο έτσι ώστε το ζήτημα να συζητηθεί σωστά και να μην το ε, συζητάμε υπό μορφή επικεφαλίδων. Τίμωθη, Ήθελα να ακούσω την Επιτροπή, αλλά μπορώ να αντιδράσω στα σχόλια. Ένα πράγμα είναι σημαντικό. Έχω ήδη λάβει πολλές γλωμοδοτήσεις, νομικές και μη. Και όπως γνωρίζει η Σάρα, οι δικηγόροι γνωμοδοτούν γνωμοδοτούν και εκφέρουν γνώμες που μπορούν να αμφισβητηθούν ή να γίνουν δεκτές ως έχουν. Εν πάση περιπτώσει δεν ε, μπορώ να λάβω τίποτα υπό απόλυτους όρους. Θα αρχίσουμε με την έκθεση αυτή, θα έχουμε κάτι διαθέσιμο το φθινόπωρο και τότε θα λάβουμε υπόψη παραμέτρους που ε, προϋπάρχουν ή όχι με βάση τα δεδομένα της στιγμής. Και αυτό θα πρέπει να γίνει δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η πρόταση αυτή είναι δεδομένη και δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε την ε, πρόταση της Επιτροπής εμείς θα βασιστούμε στη δική μας πρόταση και όχι στις Κομισιόν. Θα επανέλθουμε επί του θέματος και ελπίζω να έχουμε ε, μια καλή έκβαση. Τώρα στρέφομαι προς την Επιτροπή. Θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για τις συζητήσεις διμερώς ή ό,τι άλλο θέλετε και να σας δώσουμε τα στοιχεία που προανέφεραν οι συναδελφοί σας, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ άλλο επί του θέματος. Το Συμβούλιο. Όχι, εντάξει. Τότε θα επανέλθουμε επί του θέματος ε, αργότερα, λεπτομερέστερα. Κλείνουμε τη συνεδρίαση, λύεται η συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε με τους συντονιστές της 3 και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα αρχίσει τη συνεδρίασή της στις 3.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.